Καλημέρα σας, να αρχίσουμε παρακαλώ. We have a, our rapporteur, we have uh, one of our, our leading shadow Είναι εδώ η συγητής μας, ε, η κυρία Σουαλτεμόζα που είναι μία από τις βασικές και όθησης ηχήτριες ο κύριος Σβάπ που είναι ένας ε, ενδιαφερόμενος παρατηρητής, οπότε νομίζω είμαστε αρκετοί για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. To, um, our second second day of work this week. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Υπάρχει το πακέτο εναρμόνισης, ε, υπάρχει ε, η εσωτερική αγορά και βλέπω ότι η πιο ενθουσιώδης είναι εδώ. Και είναι εδώ ε, και ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος προφανώς είναι και εκείνος πολύ ενθουσιώδης, μια και είναι εδώ πρωί-πρωί. Είναι φίλος Επιτροπής μας και νομίζω ότι είναι εδώ και το Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Γεια σας, καλώς ήρθατε κι εσείς. Η κυρία Ρόιτοβα είναι η συγγήτριά μας για ολόκληρο το πακέτο εναρμόνισης, οπότε θα ήθελα να της δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τις ιδέες της. Έχεις το λόγο, Σουζάνα. Uh, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, την, ε, για τη συνεργασία, αλλά κυρίως τα τσεχικά θα τα πω αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια εισαγωγή για τις εννέα οδηγίες που θα μιλήσουμε, που μας απασχολούν σήμερα. Ε, είναι ένα πακέτο εναρμόνισης ε, και θα ήθελα να σας δώσω ένα πλαίσιο. Πριν από τέσσερα χρόνια ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια Σκοπός ήταν η αντικατάσταση, η αντικατάσταση ε, ορισμένων οδηγιών λόγω της ε, αγδαίας εξέλιξης στις αγορές ε, και την τεράστια αλλαγή που επέφεραν οι εισαγωγές από την Κίνα. Ήταν πολύ μεγάλες οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις και θελήσαμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δυνατότητα εποπτείας της αγοράς. Μετά από ευρεία συζήτηση, οι απαιτήσει για ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας έγιναν αυστηρότερες. Οι αλλαγές αν εγκριθούν θα έχουν ε, θετικό αντίκτυπο και στους καταναλωτές γιατί θα έχουν ε, καλύτερη ε, εξασφάλιση ότι είναι ασφαλέστερα τα προϊόντα και καλύτερων προδιαγραφών τα προϊόντα που αγοράζουν. Έχουμε λοιπόν ένα πακέτο εννέα οδηγιών που ευθυγραμμίζονται βάσει του 768 κάθετος 2008 λαμβάνουν υπόψη διάφορες ρήτρε που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προβαίνει σε νέα νομοθεσία. Είναι λοιπόν μια επιλογή οδηγιών που δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν στο άμεσο μέλλον ξανά. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχωνεύσει και να εναρμονίσει διάφορους ε, τομείς ώστε να ε, εκμεταλλευτεί την ε, καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε για την εναρμόνιση των οδηγιών αυτών. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποστήριξή μου σε σχέση με την προσπάθεια ενημέρωσης της νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα σχολιάσει άλλα ζητήματα που υπερβαίνουν το πλαίσιο της συγκεκριμένη αναδιατύπωση ε, εκτός εάν ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Να πω επίσης ότι σε γενικές γραμμές ε, το πακέτο για τα αγαθά είναι πολύ ικανοποιητικό και οι νέες οδηγίες λειτουργούν καλά στην πράξη Η μεταφορά του 768 κάθετος 2008 στο ε, πλαίσιο του πακέτου αυτού θεωρείται επιτυχής. Καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να ξαναρχίσει παλιές συζητήσεις, ε, ζητήματα που έχουν αποφασιστεί σε σχέση με ε, το πακέτο για τα αγαθά. Ήρθα εγώ σε επαφή με την Business Europe, με την Digital Europe και άλλες ενώσεις επιχειρήσεων δεν ακούσαμε ιδιαίτερα σχόλια, ούτε υπήρξαν τομεακά ζητήματα κατά τη διάρκεια της επαφής αυτές. Ήρθα και σε επαφή με καταναλωτές, με οργανισμούς καταναλωτών ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία τους ε, κατά την αναθεώρηση κάποιων λεπτομεριών. Επίσης, μαθαίνω ότι η τεχνική συζήτηση για το περιεχόμενο της οδηγίας στο Συμβούλιο θα γίνει μάλλον πριν από τον Ιούνιο αποφάσισε το Συμβούλιο να το συζητήσει με πακέτο ε, πέντε, ως πακέτο 5 οδηγιών ε, στο παράρτημα του 768 κάθετος 2008 ενώ το πιο τεχνικό κομμάτι θα συζητηθεί από, ένα ε, συγκεκριμένο, από μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας... η οποία όμως δεν έχει αρχίσει τις εργασίε της ακόμα. Μόνο τα αυστριακά σχόλια γνωρίζουμε. Υπήρξαν τρει-τέσσερι συνεδριάσεις στο Συμβούλιο μέχρι τώρα υπό την πολωνική και δανική αντιπροσωπεία και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 28 Μαρτίου θα εγκρίνει τη σχετική της νομοδότηση. Γι' αυτό λέω να το συζητήσουμε 8 Μαΐου εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και όχι στις 25 Απριλίου. Θα ήθελα να ακούσω όμως ε, κάποιες διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένα ζητήματα. Υπήρξαν και κάποιες ανησυχίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τους stakeholders. Μου εξήγησε ορισμένα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι οι σκιώδεις πρέπει να τις γνωρίζουν και εκείνοι. υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει εξωτερικών φορέων με τι οποίε δεν συμφωνώ απολύτω, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν και εκείνοι στη διαβούλευση. Η Διεθνής Ένωση Ερασιτεχνών του Ραδιοφώνου μας είπαν ότι αντιμετωπίζουν ορισμένα, έχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις συχνότητες ε, ε, στο ραδιοφάσμα και γνωρίζω ότι υπάρχει μια εξαίρεση σχετικά με το θέμα αυτό στην οδηγία, αλλά όχι στην τρέχουσα εκδοχή της. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση μιας ε, ενιαίας δήλωσης συμμόρφωσης. Το θέμα είναι θα πρέπει να είναι μία για όλες τις οδηγίες ή αν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις ε, για κάθε μεμονωμένη οδηγία. Υπάρχουν επιχειρήματα κατά αυτού ότι για παράδειγμα υπάρχει το κόστος της εκτύπωσης, πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς ε, οι λεπτομέρειες βάσει των ε, προτύπων ε, και υπάρχουν και ζητήματα εποπτείας από αρμόδιες αρχές σε διάφορα Η εφαρμογή το θέμα της εφαρμογής των κανόνων για αγαθά τα οποία ήδη υπάρχουν στην αγορά. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για το χαμηλό βολτάζ και πάλι τίθεται αυτό το θέμα του κόστους εκτύπωσης όπως επίσης και του ε, μεγάλου αντίκτυπου στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που η Γενική Διεύθυνση Υγείας ε, και Καταναλωτών ε, πέρασε την τελευταία στιγμή και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα έχει νόημα στην πράξη. Μία ακόμη ανησυχία του κατά πόσο θα αναφέρεται ο παραγωγός στο προϊόν. Κάποιοι κανονισμοί δίνουν τη δυνατότητα αυτής της, ε, της πλήρωσης αυτής της προϋπόθεσης ε, στα έγγραφα του προϊόντος, αν δεν είναι δυνατόν ε, να, γράφετε να αναγράφεται πάνω στο προϊόν το όνομα του παραγωγού, το θέμα είναι κατά πόσο θα έπρεπε να αναφέρεται και ο ιστότοπος του παραγωγού, για να μπορεί κανείς να τον βρει πιο εύκολα. Ένα ακόμη ζήτημα είναι το θέμα των εξυγχρονισμένων κανόνων για τον ορισμό της ασφάλειας, για την οδηγία προς χαμηλή τάση. Γιατί υπάρχουν σήμερα για την ασφάλεια αυτή στη σχετική οδηγία πολύ πιο συγκεκριμένοι ορισμοί. Και δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο για ποιο λόγο θα έπρεπε να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια των επίπλων, για παράδειγμα, από ότι για τα σίδερα. Ούτω ή άλλω είναι γνωστά τα πρότυπα για την ασφάλεια, που ρυθμίζουν την ασφάλεια, αλλά θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο αυτές οι απαιτήσει δεν έχουν ε, ε, συμπεριληφθεί απευθείας στο κείμενο της οδηγίας. Ένα ακόμη πρόβλημα που έχουμε, το οποίο εντόπισε το Συμβούλιο, αφορά τις εταιρείε που εγκαθιστούν ανελκυστήρες. Θα έχουν ευθύνη σαν να ήταν παραγωγή. Και αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Επίση, υπάρχουν κάποιες ανησυχίε για την ασαφή εναρμόνιση των προτύπων. Για άτομα με ειδικέ ανάγκες που τους είναι δύσκολο να μπουν σε έναν ελκυστήρα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο σαφής η ερμηνεία στο κείμενο της οδηγίας. Και δεν καταλαβαίνω γιατί στην απόφαση 768 2008 για τα, για, για τα μέσα, για τα, τις μέτρησης ζητήθηκε να συμπεριληφθούν ε, λεπτομέρειες ε, για τους ε, αγοραστές και τους προμηθευτές για 10 χρόνια. Μεγάλο αυτό το διοικητικό άχθος και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Και για το άρθρο 14 θα ήθελα διευκρινήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο ορισμός των όσων αναφέρεται εκεί. Όσον αφορά επίσης την ανεξαρτησία της ε, εταιρείας ε, κοινοποίησης, θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τις ε, μη αυτόματες, τα μη αυτόματα όργανα ζήγησης, δεν καλύπτεται το θέμα της ασφάλειας των καταναλωτών και θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα βασικά όργανα για ειδική χρήση και για μη ειδική χρήση και μιλάω για το άρθρο 6 της οδηγίας γιατί μια, ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν προκύπτει από την απόφαση. Πέρα όμως από την απόφαση, στις διάφορες οδηγίες υπάρχουν διάφοροι κανόνες ε, ε, προσφυγής ε, από διάφορους φορείς και προβλέπονται κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο. Από τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχουν νέα, νέοι κανόνες για κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κανονικά τέτοιου είδους κανόνες δεν θα έπρεπε να δημιουργούν προβλήματα στο μέλλον. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα που εντόπισε το Συμβούλιο για τα προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα και πρότεινε μία, ένα κείμενο βάσει του οποίου οι απαιτήσει που αναφέρονται στην οδηγία πρέπει να αναθεωρηθούν. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό για την ε, εποπτική αρχή. Αν αφορά, ας πούμε, ένα τμήμα του προϊόντος μόνο. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή οι όροι. Πρέπει να εναρμονιστούν ή όχι. Θα ήθελα να υπάρξει ένα πιο σαφής ορισμός για την υποχρέωση του αριθμού ε, ταυτοποίησης στη δήλωση ε, συμμόρφωσης. Μιλάω για την υποχρέωση αναφοράς δεδομένων πάνω στο προϊόν. Από ό,τι κατάλαβα, τα πράγματα δεν αλλάζουν σε σχέση με τις τρέχουσες οδηγίες, απλώς μεταφέρονται σε ένα διαφορετικό σημείο πριν από τη σήμανση ε, CE, Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πρώτα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μετά ο εισαγωγέας και μετά ο διανομέας. Μιλάω για το σημείο F για τις απαιτήσει ασφάλειες, για τη γενική ασφάλεια. Και θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μου να συνεργαστώ με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τους οποίους θα ήθελα να συναντήσω τον Απρίλιο, το αργότερο, και ευχαρίστω να ακούσω όλα τα σχόλια και όλες τις ιδέες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουμε το κείμενο των οδηγιών σε σχέση με τα 12 αυτά σημεία που ανέφερα σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ακούσω βέβαια και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί θα είναι δύσκολο και για εκείνους να μας πούν εδώ όλες τις λεπτομέρειες ε, αλλά για τα διαδικαστικά οι οδηγίες υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αναθεώρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει όμως να τροποποιήσει μόνο τα σημεία τα οποία αναφέρονται, ε, τονίζονται στο κείμενο. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποσύρει τις προτάσεις αν υπάρχουν σοβαρές αλλαγές. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, η απόφαση 768 ε, του 2008 ισχύει και εκτός από κάποιες μικρές διαφορές ή ε, προσθήκες δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σημαίνει ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ελάχιστος Το θέμα είναι, μπορεί να δεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδυναμώνεται ο ρόλος του σε τέτοιο βαθμό. Γιατί σε ορισμένες αιτιολογημένες περιπτώσεις θα μπορούσε να προβεί σε σοβαρές αλλαγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Ευχαριστώ, Σουζάννα Ροίτεβα. Πολύ δύσκολο και περίπλοκο έργο ανέλαβες και το διεκπαιρέωσες εξωτικά θα είναι πολύτιμο να δεμηνηθούν στους και στα διάφορα σημεία. Ξέρω ότι τα έχεις ε, σημειώσει προσεκτικά εκεί. Και θα καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια πρώτη απάντηση. Και θα συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα προς το τέλος. Είπε ότι ήθελες περισσότερο χρόνο στο, εν το μέσο του χρονοδιαγράμματος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Κρότσμαν, όχι. Η κυρία Ρούλα είναι εδώ. Άσλεϊ Φόξ έστειλε σημείωμα, το οποίο θα παρουσιάσω, και ο κύριος Σφάμπ. Ο κύριος Η κυρία Σαλεμόζα πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κυρία Ρόιτοβα, για την παρουσίαση, για το όλο πακέτο. Είναι μεγάλη δέσμη μέτρων. Θεωρώ σημαντικό ότι εξετάζουμε σοβαρά το θέμα το όλο νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικότατο. Τα αγαθά στην εσωτερική αγορά θέλουμε να είναι ασφαλή. Θέλουμε να έχουμε καλή υποπτία της αγοράς που λειτουργεί σωστά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στις νέα οδηγίες μαζί. Πρέπει να θυγραμμίσουμε όλες τις οδηγίες με το περιεχόμενο της απόφασης σαν Πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο να μην προβλέψουμε λιγότερες υποχρεώσεις για τους εμπορευομένους από αυτές που προβλέπονται στην 768. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιγράψουμε λίγο πολύ το κείμενο της 768. Να μην το αλλάξουμε. Είναι σημαντικό για μένα να είναι συνεκτικό το σύστημα και οι υποχρεώσεις να είναι ίδιες για όλους τους εμπορευομένους. Έτσι θα είναι πιο εύκολη η υποπτία της αγοράς του πλευράς αρχών και θα λειτουργεί σωστά η υποπτία. Ευχαριστώ που εισάκουσες τις διάφορες στοιχές που εμπεριέχουν τις διάφορες οδηγίες. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Ίσως σε κάποιες οδηγίες να κάνουμε μικροαλλαγές. Σε συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Για μένα και την ομάδα των σοσιαλιστών είναι σημαντικότατο να μην αλλάξουμε τίποτα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι εμπορευόμενοι, όσον αφορά ανιχνευσιμότητα, εποπτεία αγοράς κλπ. Άποψή μου, 768 να αντιγραφεί στις οδηγίες. Και μετά στις λεπτομέρειες των άλλων οδηγιών κουβεντιάζουμε. Έθεσε στο θέμα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο όλο θέμα επειδή ο ρόλος μας είναι μικρός. Θα ήταν χρήσιμη μια συζήτηση περί αυτού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει το έργο μας εδώ όμως, αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να ασχολούμεθα με το πακέτο αυθυγράμμισης... και ίσως τους συντονιστές και εδώ ίσως να συζητήσουμε εκτενέστερα ποιος θα είναι ο ρόλος μας σε αυτές τις αναθεωρήσεις. Ίσως να είναι γενικότερο το πρόβλημα και όχι όσον αφορά το συγκεκριμένο πακέτο. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε γρήγορα καλές λύσεις. Θα συναντηθούμε, καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε όλα αυτά λεπτομερώς. Είναι αρκετά τεχνικό το θέμα. Και ίσως να είναι δύσκολο οι άλλοι να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις. Ας συναντηθούμε και ας το κουβεντιάσουμε. Υποστηρίζω όμως ταχεία προσέγγιση. να κρατήσουμε μαζί και τι εννιά οδηγίες και να αντιγράψουμε λίγο πολύ την απόφαση. Διότι, διότι υπήρξε μακρά και καλή συνεργασία το 2007 και 2008 στο πακέτο για τα αγαθά που συζητήσαμε εκτενώς τι υποχρεώσεις πρέπει να προβλέπονται για τους εμπορικούς εμπλεκομένους. Οπότε το Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί εργασίες και δημοκρατικός πώς είναι καλό να αντιγράψουμε όλα αυτά στις νέες οδηγίες. Και προσβλέπω στο μελλοντικό μας έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπες. Θα σχολιάσω αργότερα. Αλλά ως εισηγήτρια για τις γενικότερε οδηγίες και επειδή εμείς είμαστε θεματοφύλακες στο πακέτο των αγαθών, σωστά μας τα Και έχουμε και την αναθεώρηση οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων που επίκειται. Γι' αυτό παρακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Πρέπει εν τω μεταξύ να προωθήσουμε το πακέτο τη κυρία Ρόιτεβα. Κυρία Ρούλε. Και εγώ τι θα πρέπει να πω για το πακέτο για να, την ανάπτυξη μιας κοινή γλώσσας, όλες αυτές οι οδηγίες να ισχύουν σε ένα κοινό πλαίσιο, ένας κοινό ορισμός και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτό, διότι πάλι θα δημιουργηθεί σύγχυση αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το βρίσκω σωστό να παραμείνουμε σε αυτό το πακέτο και να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα και τους όρους, που, ορολογίες που χρησιμοποιούνται. Για το ρόλο του Κοινοβουλίου το κατανοώ κυρία Ρόιτοβα. Σε αυτό τον τομέα είναι σχετικά περιορισμένος ο ρόλος της Ευρωβουλής. Από την άλλη πλευρά έχει η κυρία Μόζε απόλυτα δίκαιο και ο κύριος Μάκομ Χάμπερ όταν κάνουν λόγο για την εξέταση του πακέτου και αυτό θα γίνει στο μέλλον. Τότε θα έχει ένα ρόλο που θα διαδραματίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε συμφωνηθεί για το πακέτο αυτό όταν ε, πρόκειτο να γίνει ότι την οδηγία ουσιαστικά θα την ευθυγραμμίζαμε να συμμορφωθεί, να προσαρμοστεί και αυτό είναι ακριβώς η δουλειά της έκθεσής σας, αυτή η ευθυγράμμιση. Έχετε πλήρη υποστήριξη από μας και φυσικά πρέπει να συζητήσουμε θέματα τα οποία αναφύονται, αλλά δεν πρέπει να παρακλίνουμε από το ότι κοινού όρους και ορολογίες θα χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ. Uh, well, αν μιλήσω εκ μέρους του Άσλι Φόξ και αυτός παρακολουθούσε το θέμα εκ του και θα στείλω και σημείωμα και στην Σουζάνα. Νομίζω, τονίζοντας αυτά που είπα προηγουμένως, μετά από αυτά που είπε η κυρία Σόντερ Μόζε, υπάρχουν σαφείς απαιτήσει για όλους τους εμπλεκομένους, για τα καθήκατα των διαφόρων εισαγωγέων, των κατασκευαστών και άλλων φορέων πρέπει να υπακούν σε συγκεκριμένε προ... απαιτήσει. Και είναι και ο ρόλο των εποπτικών αρχών που καθορίζεται επακριβώ. Διότι δηλαδή είναι από τα θέματα τα οποία συνεχώ εξετάζαμε ήταν το θέμα τη εποπτεία των αγορών, που θα πρέπει να διενεργείται με συνέπεια σε ψηλά επίπεδα. Συνεχώ. Όλα αυτά κρύβονται πίσω από την πρόταση. Και πήραμε και την ανάλυση συνεπιών. Εκεί είδαμε ότι δεν πρόκειται περί του περιεχομένου, περί διοικητικών ε, διαδικασιών πρόκειται και με το σεβαστούμε. Αυτό κατά την άποψή μου δεν μειώνει, την άποψη, δεν μειώνει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Έχουμε συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουμε καθορίζοντα το πλαίσιο και στι ευρύτερε δημόσιε πολιτικέ και τα θέματα δημόσια ασφάλεια. Ασφάλεια του κοινού, μάλλον. Και γι' αυτό προβλέπω τι σχετικέ διατάξει. Ασχολούμαστε με το θέμα τώρα και στο μέλλον στην αναθεώρηση της οδηγίας περί προϊόντων. Άρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κυρία Ρόιτοβα αναφέρθηκε σε κάποια λεπτομερή ζητήματα. Αυτά προβληματίζουν και τον κύριο Φόξ. Εκαλύφθηκε ο Φόξ από αυτά που είπε η κυρία Ρόιτοβα. Και για τα διάφορα σήματα πια ενδείκνυνται για να επιτευχθούν οι στόχοι για να είναι ασφαλέστερα τα προϊόντα ή πώς αντιμετωπίζονται τα ανασφαλή προϊόντα. Όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης, τίθεται θέμα εδώ αν χρειάζεται υποχρεωτική απέτηση για ενία δήλωση που θα καλύπτει όλες τις κοινωτικές πράξεις, αν κατασκευαστής παράγει σε διαφορετικούς τομείς. Θεωρώ ότι θα μπορεί να αποφασίζει ο κατασκευαστής πώς θα το αντιμετωπίζει διότι μπορεί να έχει διάφορα ανταλλακτικά σε ένα φάσμα προϊόντων ή διαφορετικά προϊόντα. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ περιοριστικοί, φτάνει να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Θα σας στείλω την έκθεση του κυρίου Φόξ και θέλει να συνεργαστεί μαζί σας και να συμμετάσχει στις συνεδρίες των σκιωδών. Ο κύριος Σφάμπ κάτι ήθελε να πει και μετά ο κύριος Μακμίλαν. okay, first, Λοιπόν, μεταμορφωθήκατε τώρα εις σκιώδην. Uh, Θα do Θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Διάλογος εκτός μικρόφωνου. Οι σκιές προηγούνται λοιπόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω ένα σύντομο έγγραφο, σημείωμα του κυρίου Μάντα που είναι σκιώδη εισηγητής και κάποιε λίγε παρατηρήσει, θέλω να κάνω. Αυτή η ευθυγράμμιση στην οδηγία εναρμονισμού θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ καλό και υπό το πλαίσιο της νομοθεσίας στην οποία εργαστήκαμε. Συμφωνεί ο κ. Μάντας με την Επιτροπή ότι η ευθυγράμμιση θα είναι σημαντική συνεισφορά για τον πολιτικό στόχο μιας καλής λειτουργού, καλώς λειτουργούσας αγοράς για τους επαγγελματίες και τους οικονομικά εμπλεκόμενους ε, για να υπάρχει σαφήνεια εδώ θα πρέπει το, ε, αναδιατύπωση αυτή να συνεισφέρει, υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση ο κ. Μάντα. Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών είναι ορόσημο ακρογωνίω λίθο στην αγορά και βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά της ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Νομοθετικές απαιτήσει για αγαθά είναι όλο και πιο περίπλοκα θέματα για τους νομοθέτες, όλο και πιο τεχνικού χαρακτήρα και εδώ σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Σάντε Μόζερ. Καλή επιτήρηση, πολύ καλή εποπτεία της αγοράς. Χρειαζόμαστε τέτοιους κανονισμούς, αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε εποπτεία στην αγορά. Χρειαζόμαστε κανόνες και κανονισμούς, ε, ρυθμίσεις, εκθέσεις, ε, αξιολογήσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτό. Και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αυτό τώρα θα έχει ο κύριος Σβάμπ να μιλήσει για τα τελευταία λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είσαστε πράγματι σκιά της σκιά σήμερα. Ο κύριος Σβάμπ λοιπόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καθώς έχω 10 ολόκληρα λεπτά από τον κύριο Κρόισμαν, θα τα χρησιμοποιήσω πλήρως. Αγαπητέ πρόεδρε, Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική παρουσίαση της αφετηρίας ε, των πραγμάτων υπό την δική της άποψη και πραγματικά έχουμε ένα σημαντικό πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει ως Ευρωκοινοβούλιο όταν εγκρίναμε το Goods Package, την δέσμη μέτρων που συνάδελφος Αλεξάνδρ Στούμπ από τη δική μας ομάδα σημαντικά συνεισέφερε. Αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει τότε στρατηγικά θα πρέπει να τα τηρήσουμε κάπως και γι' αυτό το σχόλιο μου θα ήθελα να το θέσω καταρχήν σε δύο άξονες. Πρώτον, πρόκειται για την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004-2008 όπου οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβάσεις ε, υπό το πρίσμα μου δεν ε, πρέπει να αναδιατυπώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν είναι σωστό. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την παλιά ορολογία που είχαμε. Και θέτω αυτό το ερώτημα. Έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάτι τέτοιο. Και από τον κύριο Μακμίλαν θα ήθελα να αποσαφινιστεί στη συνέχεια αυτό. Δεύτερον, συμβαίνει το εξή. Στην οδηγία για τη χαμηλή τάση έχουμε τώρα και είναι ο μόνος τομέας που υπάρχει και η κυρία Σάντε Μόζε και η κυρία Ρούιλε το προανέφεραν και είπαν ότι σαφώς πρέπει να διατηρηθεί η ενιαία μορφή, η ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών. Μόνο που στην πρόταση για τη χαμηλή τάση ζητείται με την Declaration of Conformity, με την ε, δήλωση συμβατότητας, να υπάρχει και φωτογραφία του προϊόντος το οποίο θα, ε, η οποία θα συνάπτεται. Αυτό δεν είναι ε, κάτι λειτουργικό και είναι τα μόνα σημεία αυτά τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτεβα το έθεσε αυτό προηγουμένω. Άρα όλοι λοιπόν καλύπτονται από το ίδιο. Μα Μίλα, θα σου δώσω το λόγο. Δεν καλωσόρισα την κυρία Κέτι Ντέιβι Λάσκαρτ, που είναι πρόεδρο τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου. σω και αυτή θα ήθελα να μα πει εν συντομία πώ εξετάζει το θέμα το Συμβούλιο. Ζακ, όμω, με τα χαρά να σε καλέσω να σχολιάσει τα όσα άκουσε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την κυρία Ρόιτοβα που έκανε αυτή την εισαγωγή. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την ταχύτητα της ομιλίας σας. Δεν μπορώ να τα σημειώσω όλα. Τα δάχτυλά μου ήταν αρκετά γρήγορα να τα δαχτυλογραφήσω όλα. Και δεν έχω και χρόνο να απαντήσω και όλες τις ερωτήσεις. Γιατί μόνο πέντε λεπτά μου απομένουν. Καλωσορίζω τα σχόλια που ακούστηκαν. Κάποια από τα θέματα που ανέφερε η κυρία Ρόιτεβα είναι ζητήματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο ή που τα ακούσαμε από διάφορους ε, ενδιαφερομένους. Με τα χαράς βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει το όλο πακέτο και την αναδιατύπωση, τη διαδικασία αδιατύπωσης. Δεν θεωρούμε ότι μειοποιείται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι αυτό αποτελεί απλώς συνέχεια, έτσι το βλέπουμε εμείς, συνέχεια του πακέτου για τα αγαθά, είναι το κομμάτι της ε, εφαρμογής και ελπίζω ότι αν σωστά εφαρμόσουμε το πακέτο αυτό για την υλοποίηση δεν θα έχετε πολλά να κάνετε διότι θα κάνουμε αυτό που μας είπα να κάνουμε το 2008. Οπότε ελπίζω ότι δεν θα έχετε πολλή δουλειά γιατί απλώς θα έχουμε κάνει καλά εμείς τη δουλειά μας. Υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα και ερωτήματα κάποια λεπτομερέστερα από τα υπόλοιπα. Το θέμα της ενιαίας δήλωσης συμμόρφωσης. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ο 2008 το προτείναμε αυτό. Θεωρήσαμε ότι όταν ένας κατασκευαστής καλύπτεται από διάφορες οδηγίες, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ευκολότερο για εκείνο να έχει μία δήλωση συμμόρφωσης για να δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις διάφορες οδηγίες που αφορούν το προϊόν του και σημαντικότερο ε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τις εποπτικές αρχές. Διότι αν εμπίπτει σε έξι ή επτά οδηγίες ένα προϊόν, όπως συμβαίνει, οι εποπτικές αρχές πρέπει να ζητήσουν 6-7 δηλώσεις συμμόρφωσης. Έχουν την πλήρη εικόνα νέου. Ναι, ο μόνος τρόπος που μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο έχει τη σωστή εικόνα ο κατασκευαστής είναι διότι σε μία δήλωση συμμόρφωσης παρουσιάζει την όλη εικόνα και βλέπει κανείς κατά πόσο υπάρχει κάποιο στοιχείο που λείπει. Κατά την άποψή μας, έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε την ενιαία δήλωση συμμόρφωσης. Δικητικός πώς ίσως να δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η λογική που κρύβεται πίσω από την ενιαία δήλωση συμμόρφωσης. Και γι' αυτό για την ώρα θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την προσέγγιση. Και μάλιστα διότι συμφωνεί με αυτά που αποφασίστηκαν το 2008. Τώρα, το θέμα της ασπρόμαυρης εικόνας που γίνεται έγχρωμη, εντάξει, καλό το αίτημα για έγχρωμες φωτογραφίες. Πέρα το ότι είναι πιο δαπανηρό να έχει κανείς ασπρόμαυρη φωτογραφία από ότι έγχρωμη, ή τα πάντα είναι έγχρωμα σήμερα. Άρα χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο για να έχεις πρόβλημα φωτογραφία. Για κάποια προϊόντα μπορεί να κάνει τη διαφορά όμως. Μπορεί να κάνει τη διαφορά. Διότι βλέπεις καλύτερα το προϊόν από ότι σε ασπρόμαυρη. Τέλος πάντων. Αν αυτό είναι το τελευταίο σημείο το οποίο θα πρέπει να πολεμήσουμε, εντάξει, νομίζω θα συμφωνήσουμε, αν εκεί κολλήσουμε. Το θέμα της ταυτοποίησης του κατασκευαστού είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντα λέγαμε ότι υπάρχει κάποια ιεράρχηση. Πρώτα στο προϊόν πρέπει να μπαίνει η δεμή στα έγγραφα, η δεμή στη συσκευασία. Αυτή είναι η ιεραρχία που ακολουθούμε. Ξέρουμε ότι για πολλά προϊόντα δεν μπορεί να μπει το όνομα του κατασκευαστού στο προϊόν. Δεν θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Το θέμα της διευθύνσεως της ιστοσελίδας είναι κάτι που ανακύπτει συχνά. Εγώ θα μπορούσα να δεχτώ τη διεύθυνση της σελίδας αν κάποιος θα μπορούσε να μου εγγυηθεί ότι η διεύθυνση της σελίδας είναι σωστή και ότι προστατεύεται κατά παραπίσεις και δεν μου δεν με παραπλανεί κάποιος μέσω κάποιου προγράμματος ε, κακεντρεχούς να βγω σε άλλη στο σελίδα. Τώρα οι καταστάτες ανελκυστήρων. Αυτό είναι σημαντικό. Τι εντοπίσαμε. Τελικά, οι περισσότεροι ενελκυστήρες που τοποθετούνται σε κτίρια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εκτός της, ε, του, της σύραγγας του ενελκυστήρα, εκτός του κτίριου. Και συναρμολογούνται και τοποθετούνται εντός του κτίριου. Αναφερόμαστε στην ασφαλή χρήση των ανελκυστήρων να είναι ένα ανερκιστήρα, ο οποίο είναι ασφαλή αυτός που διατίθεται. Όμως η σημαντικότερη μάλλον φάση είναι η εγκατάσταση αυτού. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τον εγκαταστάτη και να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι εξίσου σημαντικός όπως ο κατασκευαστής των διαφόρων κομματιών των ελκυστήρα. Αν είναι σωστός, αν τα πάει καλά, αν είναι σωστά τα κομμάτια, είναι καλό, αλλά αν κάνει λάθο ο εγκαταστάτη, δεν είναι καλά τα πράγματα. Άρα και ο εγκαταστάτη πρέπει να έχει τι ίδιε υποχρεώσει όπω ο κατασκευαστή των διαφόρων κομματιών των ελκυστήρα. Δεν κάνει διαφορά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει αυτό. Οι περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει θα εγκαθιστούν ανελκυστήρε ούτω ή άλλω. Δεν θα σχεδιάζουν ούτε θα κατασκευάζουν του ανελκυστήρε. Θα συναρμολογούν του ανελκυστήρε. Άρα, δεν είναι θέμα μεγέθου επιχειρήσεω, αλλά θέμα του ποιο κάνει το τελευταίο σφάλμα που είναι και το σημαντικό. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Τώρα στα λεπτομερέστερα ζητήματα θα πρέπει να εξετάσουμε τον κατάλογο με την κυρία Ρόιτεβα. Αυτά είναι τα σημαντικά σημεία που θεώρησα ότι έπρεπε να παρουσιάσω τώρα στην πρωινή συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, που ήρθατε. α, κάτι άλλο, κάτι άλλο, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ήξερα ότι κάτι μου έλειπε, κάτι που θα αναφέρω. Ήθελα να μιλήσω για τη διαδικασία εποπτείας της αγοράς. Τι λέει το άρθρο. Ότι οι αρχές οι εποπτικές θα πρέπει να εξετάζουν όλα, όλους τους κινδύνους που παρουσιάζει, που μπορούσε να δημιουργήσει ένα προϊόν. Η διατύπωση της 768 είναι ένα απομεινάρι του διαχωρισμού κανονισμού και απόφασης και αρχικά ποιο ήταν το νόημα και ποιο είναι πιστεύουμε ακόμα το νόημα ότι η εποπτική αρχή που εποπτεύει τις αγορές όταν έχει αμφιβολία για ένα προϊόν πριν το επιστρέψει στον κατασκευαστή για διορθωτικές δράσεις θέλει να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν άλλες αμφιβολίες σχετικά με το ίδιο προϊόν ούτως ώστε ο κατασκευαστής να μην πρέπει να περάσει την ίδια δικασία επανειλημμένα. Αυτό είναι ο στόχος της διατύπωσης. Το ότι η απόφαση έχει διαχωριστεί από τον κανονισμό δημιουργεί την εντύπωση ότι λέγεται κάτι διαφορετικό. Αλλά κατά εμείς πιστεύουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τον έλεγχο που διεξάγουν οι υποπτικές αρχές. Δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα και οι διορθωτικές Δράσει κοινοποιούνται με τη μία. Να, τα κάνει, να κάνει όλες τις διορθώσεις με τη μία ο κατασκευαστή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Όπω είπε η κυρία Ρότεβα, έχουμε πάρα πολλέ λεπτομέρειε να ρυθμίσουμε. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και να γλιστρήσουμε ήρεμα προ την ψηφοφορία. Ναι, Ζακ. Όπω έλεγε η Σουζάννα Ρόιτεβα, θα συναντηθείτε με τους Κιώδης για να εξετάσετε τι λεπτομέρειε και είμαι σίγουρο ότι θα επιληθούν. Ε, κύριε Ντέιβιντ, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτή τη φάση. Όχι. Θα τα πούμε σε άλλη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Σουζάνα, να αναφέρω το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το σωστό. Νομίζω ότι προτείνεις κάποιες αλλαγές, όπως προανέφερες. Αλλά όχι αλλαγή όσον αφορά την τελική ψηφοφορία. Θα μας στείλει μεταφρασμένη έκθεση στις 11 Απριλίου. Το σχέδιο εκθέσης ζητηθεί 8 Μαΐου, προθεσμία για τροπολογίες 16 Μαΐου, συζήτηση τροπολογιών 20 Ιουνίου, ψηφοφορία 10 Ιουλίου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο και ελπίζω ότι αυτό θα ταιριάζει και με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου και αν χρειαστεί θα συζητήσουμε και με το Συμβούλιο. Διότι σε κάποια φάση το Συμβούλιο και εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπω να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πώς σας εξαρτάται όμως αυτή η διαπίστωση. Καλώς θα προχωρήσουμε και θα πάμε στη ψηφοφορία. Έχουμε δύο ψηφοφορίες, μάλλον τρεις ψηφοφορίες να κάνουμε. Διότι μετά από τις συζητήσεις τις θεσινέ όσον αφορά τα δίτροχα με κινητήρες και με μοτοσυκλέτες. Ο κ. Βάντερ Κάπταν συγητής. Ξέρουμε ότι στου Σκιώδης συζητήσατε το θέμα και θέλατε να ζητήσετε εντολή. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βάντερ Κάμπ για να μας καθαρίσει ακριβώς τι υπόθηκε και τι έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σωστά νομίζω τα συνοψίσατε. Εχθές εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολόγηση επιπτώσεων. Έχουμε μια επαρκή βάση έτσι ως θεμέλιο για να ξεκινήσουμε με τον άτυπο τριμερή διάλογο τώρα. Εδώ σε αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια εντολή από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, διότι με του σκιώδει εισηγητές θα ήθελα από πλευρά μου να ολοκληρώσουμε με θετικό τρόπο. Θέλω να τηρήσουμε την προθεσμία όπω και για τον κανονισμό. Πρόκειται για πολλέ συμφωνίε και προτάσει για το, το ίδιο, τα ίδια κεφάλαια και από πλευρά χρόνου και από πλευρά διεργασιών θα έπρεπε να βαίνουν εκ παραλίλου αυτά. Well, I I put... Μάλιστα, ευχαριστώ. Μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό προ έγκριση. Όσοι είναι υπέρ του να δοθεί εντολή προ την Επιτροπή κατά εντάξει εγκρίθηκε, σαφώς έγινε δεκτή, χρειαζόμαστε πάνω από 19 ψήφους, είχαμε ούτως ή άλλως πάνω σαφές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εντολή και θα δούμε πώς θα προχωρήσετε. Ας προχωρήσουμε στην έκθεση του κυρίου Κρόσμα τώρα για τον κανονισμό που αφορά ε, την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και τα τελωνία. Θα, δώσει, θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή για εισαγωγή πρώτα Διαρωτώ με, θα μπορούσατε να πείτε κάτι για κάποιους τομείς παιδεία τροπολογιών όπου έχουμε κάποιες δυσκολίες λόγω της διευρυμένης συνεργασίας που έχουμε με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σίγουρα έχουμε εξετάσει και τα έχουμε δει αυτά και κάποιες από τις τροπολογίες πρέπει να περάσουν και να μπορέσουν να ε, εγκριθούν χωρίς αλλαγές. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σχεώδεις εισηγητές. Είχαμε πραγματικά μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, επικοδομητικέ συζητήσει σε δύο γύρου και άκουσα επίση ότι δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία για όλε τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ελπίζω όμω ότι θα έχουμε καλές ψηφοφορίες. Ε, ευχαριστώ για την υποστήριξή σα, Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με τι ψηφοφορίε τώρα. Ευχαριστώ. Right. Ε, Εντάξει, νέο Πρόεδρο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες μας ε, για την ψηφοφορία και θα μου λένε κύριε η κυρία αν πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος ή όχι, ούτως ή άλλως θα το δούμε αυτό και για θέματα τα οποία έχουν, έχετε στον πίνακα ψηφοφορίας στο τροπολογία 110 τώρα, υπέρ, κατά, α, απορρίφθηκε σαφώς, 15 για διαγραφή του κυρίου Κρόισμαν υπέρ, κατά, α, α, και αυτή απορρίφθηκε, η 113 υπέρ, κατά απορρίφθηκε. Η 112 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 112. Uh, is... ψηφοφορίας απορρίφθηκε σαφές το αποτέλεσμα. Τώρα, διεθνέ εμπόριο εγκρίθηκε υπό τον κανονισμό 50, το άρθρο του κανονισμού 50 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όλε οι υπόλοιπε 111, 114, 115, 16 και 18 καταπίπτουν και έτσι περνάμε στην τροπολογία 119 έγκστρομ, υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 120 υπέρ κατά απορρίφθηκε 121 υπέρ κατά Εγκρίθηκε σαφές το αποτέλεσμα. 122 υπέρ κατά απορρίφθηκε η 123 η 124 και η 10 από κοινού άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών παρακαλώ Πέρα ψηφοφορία τώρα απορρίφθηκαν η 125 αποσύρθηκε της νομικών υποθέσεων 11 τώρα θεωρείται ότι εγκρίθηκε υπό τον κανόνα 50, υπό το άρθρο 50 του κανονισμού η 131, η 127, η 130, 132 όλες καταπίπτουν η 126 129, 128 και 133 έχουν αποσυρθεί, 135 και αυτή καταπίπτει. Και έτσι πάμε κατευθείαν κάτω στην 141 τροπολογία. Έγκστρομ, παρακαλώ. 141 Έγκστρομ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. The vote is... Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 140. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 140. The vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Έτσι 139 και τις νομικών υποθέσεων 12 καταπίπτουν. Τροπολογία 144, Μακλάρκιν, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Η 142, Σαλβίνη, Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε την 142 Σαλβίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Oh, sorry, that's uh, I think The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε, είναι σαφές. Δεν είχαμε σαφές ε, μήνυμα. 143 της κυρίας Χέντ, υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίθηκε. Και έτσι Έχουμε την ΙΝΤΑ 9 που είναι συμβατή με την 143 του Διεθνούς Εμπορίου 9. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Την 9 τροπολογία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Είναι σαφές. Και τώρα η τροπολογία 145 δεν είναι σαφές τι θα γίνει εδώ η 145 δεν είναι παραδεκτή γιατί ήδη καλύπτεται από άλλες. Η 146 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 147 της κυρίας Head. Όσοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίθηκε, είναι σαφές. Οι 149 και 150 ταυτόσιμες Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία 149-150. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 19 υπέρ 19 εναντίον ισοψηφία απορρίπτονται. Εν πάση περιπτώσει, πιο γρήγορα να προχωρούμε με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες γιατί δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. 151 Vice Gerber. Άρχεται η ψηφοφορία. 151. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Η 16 Κρόισμαν. υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 17 Κρόισμαν. υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Η συμβιβαστική 1 εγκρίθηκε. Και έτσι πάμε στην τροπολογία 153 της κυρίας Χέντ. υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 154. Μη παραδεκτή, ήδη καλύφθηκε. 155-156 αποσύρθηκαν και περνάμε στην 161 της κυρίας Χέντ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 161. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 163 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Η 164 δεν είναι παραδεκτή. Η 19 του κυρίου Κρόσμαν υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 165-166 υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν. Διεθνούς εμπορίου 10 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 του κ. Κρόισμαν. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Ε, Διεθνούς Εμπορίου 11. Είναι συμβατή. Είναι τα 11. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11 της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 21 του κ. Κρόισμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 21 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Έχουμε μια προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 167 που αναφέρεται στον πίνακα ψηφοφορία. Όλοι το δέχεστε, υποθέτω. Όσοι είναι υπέρ της προφορικής τροποποίηση, κατά εγκρίθηκε αυτή η προφορική τροφοποίηση Η 167 καταπίπτει, 169 τώρα υπέρ. Νομίζω ηλεκτρονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 169. Πέρας πληροφορία, εγκρίθηκε. Η 168 καταπίπτει, 170 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Νομικών υποθέσεων 13 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Νομικών υποθέσεων 14 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 171. Γκάλο. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 172. Μακλάκιν. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε σαφέ. Τροπολογία 173 και ίντα 12, Διεθνούς Εμπορίου 12. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών. 173 και ίντα 12. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκαν αυτές οι δύο τροπολογίες. Η 174 Engström. υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Η 176 Angstrom Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 176. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 177. Έγκστρομ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 178. Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 179. Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 22. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 180. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 180. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η 182. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 182. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα και αυτή εγκρίθηκε. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 183 καταπίπτει και των νομικών υποθέσεων 15 είναι συμβατή. Υπέρ της 15 γιούρι υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και έτσι πάμε τώρα κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά. Και αυτή εγκρίθηκε. Και πάμε στην 191 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 191. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Η 192 Κρόιτσμαν υπέρ κατά εγκρίθηκε. 25 καταπίπτει. 26 Κρότσμαν υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τζούρι 17 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 194. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 21 ψήφοι υπέρ, 15 εναντίον. Νομικών υποθέσεων 18 είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 27, 195, 196 και 19. Ψηφίζουμε αυτές τις τέσσερις τροπολογίες ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Έγινε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούστηκε. Εγκρίθηκαν αυτές. 197 και 198 καταπίπτουν, 199 τώρα. Τροπολογία 199 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 200 τροπολογία. 200. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την τροπολογία 200. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 201 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίθηκε. 202 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 202 πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 203 και Γιούρι 20, 20 ε, υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν Πάμε στο άρθρο 18. 205 τροπολογία και jury 21. Υπέρ αυτών των δύο. Κατά εγκρίθηκαν. Η 204 είναι συμβατή. Υπέρ της 204. Κατά και αυτή εγκρίθηκε. 206 και 207 καταπίπτουν επειδή καλύπτονται ήδη από το άρθρο 51. Ή θα ψηφίσουμε. Τι λέτε πρέπει να ψηφιστεί 207. Πρώτη υποπαράγραφος της ε, τροπολογίας Prendergast. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όσοι είναι υπέρ τη 207, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τώρα, 208, Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 28 αποσύρθηκε, 29 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 30 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 209 καταπίπτει. 210 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Η 31 αποσύρθηκε. 211 head υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 212 head υπέρ. Εγκρίθηκε. τα 14 εγκρίθηκε υπό τον κανόνα 50. Τροπολογία 32 Κρότσμαν υπέρ κατά απόχέ εγκρίθηκε τροπολογία 33 Κρότσμαν υπέρ κατά εγκρίθηκε 34 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 213 Σαλβίνη υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε και 214-215 καταπίπτουν 216 Σαλβίνη υπέρ κατά εγκρίθηκε 35 τώρα υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 218 και γιούρ 22 καταπίπτουν. 36 Κρόσμαν, υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 37 Κρόσμαν, υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 38 Κρόσμαν, υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 219 Έγκστρομ στο άρθρο 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 220. Έγκστρομ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 39. Κρόισμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 221. Σαλβίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 221. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και τώρα τροπολογία 40. Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 42 και 222 θεωρείται ότι εγκρίθηκαν επειδή συνδεόντουσαν με την τροπολογία 33 38 με τις άλλες τροπολογίες αυτές. Περνάμε στην τροπολογία 223 Σαλβίνη υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 224 καταπίπτει, 225 Σαλβίνη υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και έτσι η 226 καταπίπτει, 227 και Γιούρι 23 υπέρ αυτών εγκρίθηκαν. 228 και Τζούρι 24 υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν. 229 Σαλβίνη υπέρ κατά εγκρίθηκε. 230 καταπίπτει, 231 αποσύρθηκε, περνάμε στη 43 υπέρ. Κατά. Υπέρ τη 43. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, είναι πιο εύκολο. Ψηφίζουμε την τροπολογία 43, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 23 ψήφοι υπέρ, 17 εναντίον. Η 233 καταπίπτει. 232 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 232. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 234 αποσύρθηκε. Πάμε στη 44 Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 235 και Γιούρι 25. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών ηλεκτρονικά επ' αυτών των δύο τροπολογιών. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν αυτές οι δύο. Συμβιβασμός 4, συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά στη συμβαστική τροπολογία 4. Η 4, η συμβαστική 4 λοιπόν, εγκρίθηκε μάλιστα. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία, συμβαστική τροπολογία τώρα, Α, όχι, έχει αποσυρθεί αυτή, μάλιστα. συγγνώμη. 46 τροπολογία, υπέρ. Θα αρχίσει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 2.39 και Γιούρι 27 και η 2.38 καταπίπτουν. Τροπολογία 47 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 48 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Έτσι 2.40 καταπίπτει. 49 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία στη συμβιβαστική 6. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και περνάμε στις τροπολογίες 51 και 242. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκαν. Τροπολογία 243. 2.43. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά στην 2.43. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2.44. Head. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 245 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 52 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 246 αποσύρθηκε. 247 τώρα υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 53. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 54 τοπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 55 υπέρ. Θα ψηφίσουμε την 55 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, Εγκρίθηκε λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, εγκρίθηκε. Μάλιστα. Η 55 εγκρίθηκε, για να είμαστε σαφείς. Η 248 τώρα. Καταπίπτει η 248. Η 28 θεωρείται ότι εγκρίθηκε υπό το άρθρο 50. Η άλλη καταπίπτει, 250 αποσύρθηκε, 251 δεν είναι παραδεκτή. Περνάμε στην 56 τροπολογία, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 57 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 29. Γιούρι. Γιούρι 29. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 2.52 με την προφορική τροποποίηση του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Η 2.52 καταπίπτει. Η Γιούρι 30 καταπίπτει. Η 2.53 με την προφορική τροποποίηση τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 2.54. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 2.54. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 255 με την προφορική τροποποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 255 με προφορική τροποποίηση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε αυτή. Η 255 καταπίπτει λοιπόν. 258 Χένσλικ υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 58 εισηγητού υπέρ κατά εγκρίθηκε 259 υπέρ κατά εγκρίθηκε η 59 καταπίπτει 2.57 καταπίπτει, 2.56 καταπίπτει, τροπολογία 60 τώρα. Θα ψηφίσουμε αυτήν, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Με χαρά θα το ακούσετε αυτό. Αιτιολογική σκέψη 2. Τροπολογία 62. Έγκστρομ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 61. Τζούρι 1. Υπέρ αυτών. Κατά. Εγκρίθηκαν. Ίντα 1. Υπέρ. Να επαναλάβουμε. Υπέρ του Διεθνούς Εμπορίου. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 64 συμβατή υπέρ της 64 κατά απορρίφθηκε τροπολογία 67 υπέρ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 67 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκε τροπολογία 66 υπέρ κατά Απορρίφθηκε, είναι σαφέ. Τροπολογία 65 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 65. Πέρα ψηφοφορία τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η τροπολογία 1 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 3 υπέρ. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 3 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 73. 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Η τροπολογία 73 απλώς. Ναι. Εντάξει. Ακυρώνεται αυτό. Υπέρ. Κατά. Η 73 απορρίφθηκε. Είναι σαφέ Η 74 τώρα. Υπέρ. Κατά. Και αυτή απορρίφθηκε. Μάλιστα. 76. Η 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 76. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 75 τώρα. Υπέρ. Νομίζω θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 75. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα λοιπόν εγκρίθηκε η Jury 3 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 5 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και έτσι πάμε στην 79 και στην ΙΤΑ 2 καταπίπτουν το ίδιο και η 78 και Τζούρι 4. Πάμε στην τροπολογία 6, Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ, κατά, ναι, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 14, για διαγραφή 8, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 11 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η των νομικών υποθέσεων Jury 8 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε. Και έτσι περνάμε τώρα στην τροπολογία 101 υπέρ κατά εγκρίθηκε. τα 5, 6 και 7 εγκρίθηκαν. Ήδη συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την συμβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα αυτή η συμβαστική τροπολογία απορρίφθηκε. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο τα συστατικά τμήματα αυτής της τροπολογίας. Τροπολογία 13 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 13 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε, είναι σαφές. Η 106 τώρα. Τροπολογία 106, όσοι είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 104 της κυρίας Γκάλο. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 104. Πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 20 ψήφοι υπέρ 18 εναντίον. Η Τζούρι 9 λοιπόν καταπίπτει. 105, 105 αποσύρθηκε. Τροπολογία 14. Κρότσμαν υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 107 καταπίπτει. Η 108 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και η 109 τώρα υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και τώρα λοιπόν θα περάσουμε στην τελική ψήφιση, τελική ψηφοφορία Άρχεται η τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 36 ψήφοι υπέρ, 3 εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Κρότσμαν λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. So, thank you very much for your... Σας ευχαριστώ πολύ για την τελική σας αυτή δουλειά ως εισηγητής για την Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σας ευχαριστούσα για την εξαιρετική δουλειά σας σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την τελευταία σας αυτή έκθεση. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος στη συνέχεια να συνεχίσετε το έργο αυτό. Ίσως έχω μια πολύ καλή λύση, να είναι καλή λύση αυτή. Ευχαριστώ όλους και πρέπει να πάμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα δω αν η Ιδανική Προεδρία μπορεί να σπρώξει κάποια κράτη-μέλη. Θα δούμε αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της περίοδου. Ευχαριστώ για τα πάντα. Νομίζω ότι πήραμε πολύ καλή απόφαση σήμερα και βοηθήσουμε, βοηθάμε και τα τελωνία και τους ε, κατόχους των δικαιωμάτων. Και τα τελωνία να μειώσουμε το άχθος τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, I think we should also, um, thank you. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τις άλλες επιτροπές για τη συνεργασία τους μαζί σας. Νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση λειτουργήσε πολύ καλά. Προχωράμε. Πάμε στο, στην πληροφορία για τον προπολογισμό. Θα δώσω στον κύριο Μπουζόη, τον εισηγητή μας, το λόγο να πει μερικά πράγματα πολύ σύντομα, να ευχαριστήσω τους Κιώδης και του άλλους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή της, την γραμματεία της ΣΥΜΚΟ και το προσωπικό για τη βοήθειά τους και ας πάμε στην ψηφοφορία γιατί είναι και αργά κιόλας. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. 3. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία που αφορά την παράγραφο 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 καταπίπτει. Τροπολογία 12 καταπίπτει. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 απεσύρθη. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπουζόη και θα υπερσουστούμε αυτή τη θέση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η κυρία Ρόιτεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Εγώ θέλω να πω ότι υπερψήφισα αλλά δεν δούλευε το μηχάνημά μου. Οπότε θα ήθελα να καταγράψετε την ψήφο μου. Υπερψήφισα. Και εγώ. Okay, we will... Καλώς. Θα προσθέσουμε μία ψήφο υπέρ. Ευχαριστώ όλους σας για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ τους εισηγητές. Οπότε πάμε... Στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Επόμενο θέμα. Στα δύο σημαντικότερα θέματα πιθανότατα για αυτό το κύκλο εργασιών. Παρακαλώ όσοι αποχωρούν μετά τις ψηφοφορίες αποχωρήσουν ησύχως διότι έχουμε πολλή δουλειά όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα και τον κύριο Ζουβά για τη σκληρή δουλειά που έκαναν για να ετοιμάσουν αυτά τα έγγραφα που θα βοηθήσουν τη συζήτησή μα, Λυπούμε ότι δεν διατίθεται, σε όλες τι γλώσσες. Ετοιμάστηκαν όμω αρκετά γρήγορα και πιστεύω ότι βοηθούν σημαντικά το έργο μας. Έγινε επικοδομητική συζήτηση, πολύ επικοδομητική, για μια διευθέτηση πλήρη, για να πετύχουμε το στόχο που καθόρισαν οι Ευρωπαίοι Πρωθυπουργοί να καταλήξουμε κάποια, κάπου θετικά θέλησαν στο τέλος του έτους και οι συγγητές καταβάλουν τη δέουσα προσπάθεια και σκιώδης. Είναι κοινό το έργο όμως. Σας παρακαλώ, ησυχία. Αν θέλετε να συζητήσετε, εκτός αιθούσης. Θα καλέσω τον εισηγητή μας για το θέμα των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τον κύριο Ταραμπέλα, να παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας και θα συζητήσουμε και θα πάρετε το λόγο κύριε Ταραμπέλα. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος που θέσαμε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ απλούστευσης κανόνων και υγιεινών, και ασφαλών αν θέλετε, διαδικασιών για αυτές τις συμβάσεις, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θέλουμε να υπάρχει γενικότερη προσφυγή στη δημόσια σύμβαση δημοσίων συμβάσεων. Οι δημόσιες συμβάσεις, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Μπαρνιέ, είναι το 19% του αέπτος του εσωτερικού της Ευρώπης και εν ώψη της κρίσεως που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να εξερευνήσουμε στο μέγιστο δυνατόν το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι για να αυξήσουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και θα πρέπει να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία. Χαιρετίζω την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, πρόκειται περί καλής βάσης προβληματισμού ε, που ελπίζω ότι θα τη βελτιώσουμε μαζί για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η μέθοδος εργασίας ε, που πρότεινα και κοιόδους ηγητές σε μια προηγούμενη συνεδρίαση είναι ότι εφόσον μιλάμε για δύο ε, κατευθύνσεις ε, για να γίνουν πιο εύκολα συζητήσει και ο προβληματισμό, προτείνω να ακολουθήσουμε μία μέθοδο που ξεκίνησε η Ιδανική Προεδρία στο Συμβούλιο. Δηλαδή, να σκεφτούμε σε ομάδε θεματικέ, συστάδε θεμάτων. Ένα, δύο, πέντε και τέσσερα. Τι ομάδε αυτέ προτείνω ε, που βρίσκονται στο έγγραφο συνεδρίαση. Στην ομάδα 1 ε, είναι επιλογή αυξημένη των επιλογών. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία των διαδικασιών, γενικεύοντα τη διαπραγματευτική διαδικασία, ανταγωνιστικό διάλογο και δημιουργώντα συνεργασία για την καινοτομία. Ε, το υποστηρίζω αυτό, αλλά αυτή η ευελιξία δεν θέλω να οδηγήσει σε αδιαφάνεια και νομική ανασφάλεια αυξανόμενη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την νομική ασφάλεια. Θα ήθελα επίσης όλες οι διαδικασίες να υποβάλλονται στα ίδια κριτήρια της ανάθεσης. Δηλαδή, η καλύτερη οικονομική προσφορά να κερδίζει. Θα έπρεπε να καταργήσουμε απλούστατα την αναφορά στη χαμηλότερη τιμή και την πιο εποφελή οικονομική προσφορά. Θέλουμε να έχουμε τη βιωσιμότητα και άλλα κριτήρια και την ποιότητα να λαμβάνει υπόψη για λόγου τη βιωσιμότητα. Στα τα δύο, εξετάζουμε τη στρατηγική ε, επιλογή η πιο υποφελής οικονομική προσφορά και η βιωσιμότητα να λαμβάνονται υπόψη. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη επίσης ε, πτυχές που δίνουν υπεραξία στην προσφορά. Μία επιχείρηση που σέβεται ε, τους εργοδότες έχει περισσότερες δυνατότητες να είναι αξιοπιστή με ακροπρόθεσμα από μια ε, εταιρεία που πληρώνει τους εργαζομένους στη μαύρη δεν είναι μόνο κοινωνικό το θέμα, αλλά και θέμα οικονομική αποδοτικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η υπεργολοδία, η υπερβολική. Διότι ο να μην γίνονται πιο. είναι μεγαλύτερη κίνδυνη να μην γίνονται σεβαστοί οι όροι εργασία και άρα να μην γίνεται σωστά η δουλειά. Γι' αυτό η επιχείρηση υπεύθυνη για η ανάδοχο θα πρέπει να αναλαμβάνει και την... να συμμορφώνει την αρχή της ε, της υπευθυνότητας. Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ υπηρεσιών Α και Β, θέλω την άποψη των συναδέλφων μου. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να δημιουργηθεί μια διαδικασία ε, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά οι νομικές υπηρεσίες δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν. Ερώτημα. Η συστάδα 3 αφορά την πρόσφυγη στα, έγγραφα. Όλοι πρέπει να χαιρετήσουμε την ε, πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να μειωθεί το διοικητικό άχθος, δηλαδή η γραφειοκρατία. Σχετικά με αυτό το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο και κυρίω το παράρτημα 18 θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω για να συμπεριφθεί ο σεβασμό των περιβαλλοντικών, νομικών και κοινωνικών ρητρών. Η συστάδα 4 είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την ηλεκτρονική ε, σύναψη συμβάσεων και εδώ καλή πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργούνται πολλέ ανησυχίε και το μιλώ για ανησυχίε. Ε, το λέω γιατί συνάντησα πάνω από 40 ενδιαφερομένου πάνω σε αυτό το θέμα ε, και είναι ένα θέμα που συνέχεια αναφέρεται, ανησυχούν για την ηλεκτρονική διαδικασία και θα ήθελα ιδιαίτερα να θέσω το ερώτημα αυτό που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται. Πώς θα εξασφαλίζει την προστασία των στοιχείων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών αυτών συνάψεων δημοσίων συμβάσεων και αν ε, επιβάλλονται υπερβολικές επενδύσεις, κυρίως στις μικρές ε, επιχειρήσεις. Ε, μήπως είναι μεγάλο το οικονομικό βάρος και η μείωση του χρόνου που δίνεται στι ε, εταιρείε ίσω να είναι μια ψευδής καλή ιδέα και δεν είναι προ όφελο των πολύ μικρών εταιριών. Όσον αφορά τι προθεσμίε, εγώ θα ήμουν αντίθετο με την πρόταση αυτή, διότι δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει το σύντομο χρονικό διάστημα τη μικρή επιχειρησία. Στη στάδα 5 είναι επίση σημαντική. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλύπτεται εδώ και είναι ένα από του στόχου του σημαντικότερου αυτή τη νέα οδηγία ε, που σαφέστερα είναι η διευκόλυνση στην πρόσβασή του στι δημόσιε αυτέ ε, προμήθειε. Και συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, θα πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται και με τι εξουσίε που κάνουν την ανάθεση και να μην, βελτιώσουμε, να μην αυξήσουμε το διοικητικό άκθο. Ε, να μοιράζεται, γίνεται επιμερισμό σε παρτίδε είναι καλή ιδέα και εκείνο που υποβάλλει το αίτημα να εξηγεί είναι και αυτό που μπορεί όλου ενδιαφερομένου να του βοηθάει και θα ήταν σκόπιμο να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία κατά παρτίδε, ευνοούντας την ομαδοποίηση των διαφόρων προσφορών, αναπτύσσοντας ε, και τα κονσόρσια. Αυτό ισχύει στην Ιταλία και αλλού, πιστεύω. Η συστάδα των μέτρων 6 των προτάσεων αφορά την ομοδοποίηση τη ζήτηση. Εκεί δεν έχω τίποτα να αλλάξω εν συγκρίση με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συστάδα 7 αφορά τι άλλε απαιτήσει, τι διαδικαστικέ και ανάμεσα στι νέε απαιτήσει υπάρχει η μείωση του χρόνου που δίνει τι επιχειρήσει για να κάνουν την προσφορά του και αυτό μου δημιουργεί προβλήματα όπω προανέφερα. Ε, η συστάδα μέτρων 8 είναι υγιή ε, διαδικασία, μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση των διαδικασιών. Δεν θα πρέπει να έχει σαν συνέπεια όμω μια αύξηση ε, τη συγκρούσεω συμφερόντων ή αθέμητων συμπεριφερών. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε δυνατότητα διαφθορά στην λειτουργία αυτών των συμβάσεων έχοντα μέτρα διαφύλαξη. Η, η συστάδα 9 αφορά τη διακυβέρνηση και εκεί η πρόταση Ευρωπαϊκή Επίτροπη προβλέπει υποχρέωση στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μια εθνική αρχή ελέγχου αυτή η πρόταση δημιουργεί κάποιου φόβου κατανοητού από πλευρά των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν ελεγκτικέ αρχέ και δεν ήταν πρακτικότερο να του αναθέσουμε τα προβλεπόμενα καθήκοντα και ο στόχο θα πρέπει να είναι απλούστευση μέγιστη και όχι να δημιουργήσουμε νέε δομέ που θα, ε, θα αυξήσουν το διοικητικό άκθο. Μετά, στάδα μέτρων 10 αφορά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογή. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να εφαρμόσει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη ε, συνεργασία των δημόσιο τομέα, δημοσίου-δημοσίου. Προσπαθήσαμε να λύσουμε κάποια προβλήματα αν ήταν πολύ περιοριστικό ορισμό τη συνεργασία δημοσίου-δημοσίου τομέα που θα μπορούσε να εμποδίσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε περιορισμένο βαθμό όσον αφορά την κοινωνική στέγαση, παραδείγματο χάρη, όσον αφορά τα όρια. Θα ήθελα και εδώ να ξέρω ποια είναι η άποψη του συναδέλφου μου, δεν μπόρεσα εκ των προτέρων να κάνω κάποιε αλλαγέ και τη συμφωνώ με την Πρωθυπουργική Επιτροπή. Εν γέννη, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτέ είναι κάποιε σκέψει που έχω όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό θέμα που είναι πολύ περίπλοκο. Περιμένω ανυπόμονα να ακούσω τι σκέψει και όπω είχα την ευκαιρία να το πω και στου δύο αλλά το επαναλαμβάνω στου συναδέλφου. Θέλω πραγματικά να συνεργαστώ με όλε τι πολιτικέ ομάδε, με όλου του το μόνο πράγμα το οποίο διακινδυνεύει κατά την άποψή μου είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται στο, ε, στο Κοινοβούλιο. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα, το ξέρετε, προβλέπεται στην ΙΜΚΟ ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Υπάρχουν 10 επιτροπέ πέραν τη δική μα. Εμεί είμαστε επί αρμόδια. 10 όμω έχουν επιφορτιστεί να γνωμοδοτήσουν επιτροπέ. Δεν θα το κάνουν όλε, κάποια δεν θα το κάνει. Και 7 και 8 και 9 να είναι όμω, είναι σαφέ ότι θα είναι τόσε πολλέ τροπολογίε να αντιμετωπίσουμε δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ελευθερία των βουλευτών που είμαστε και είσαστε να εκφραστούμε, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα κατά πολιτικέ ομάδε να συνεννοηθούμε για την κατάσταση των τροπολογιών, θα ήταν καλό για να μην έχουμε τεράστιο ρυθμό τροπολογιών, διότι διαφορετικά αυτό δυσκολεύει πολύ τη διαδικασία και το καθήκον μα. Αποστολή μα σε αυτό το θέμα το σημαντικό, όπω υπενθύμησατε κύριε Πρόεδρε, είναι να στείλουμε σαφέ μήνυμα, σαφέ μήνυμα το οποίο το δημιουργήσουμε μαζί, ούτως ώστε να πλουστεύσουμε πραγματικά τα πράγματα και να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι όχι μόνο να δώσουμε το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι δημόσιες συμβάσεις, αλλά θέλουμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη στην οικονομική ανάκαμψη. Κάθε θολό μήνυμα θα ήταν επιβλαβές, νομίζω. Το είπα και το επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να εμποδίσω την ελευθερία που έχουμε όλοι να καταθέσουμε τροπολογίε. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα να σα ακούσω. Well, thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας τα είπατε όλα πάρα πολύ σαφώς και είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Θα μιλήσουμε για τις διαδικασίες πιο μετά. Λοιπόν, οι σκιώδεις εισηγητές τώρα. Και ο Κλάς είναι εδώ. Θα πρέπει να περιμένετε λιγάκι. Είδατε όμως ε, το έγγραφο ε, εργασίας, οπότε φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί. Μπορεί να χρειαστεί να βιαστούμε λίγο, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης μετά. Οπότε, εδώ ο Άγγελο ο κ. Κατζημαρκάκης. Ε, γεια σας. Έχετε και καινούριο ρόλο στην Επιτροπή μας. Η κυρία Ρούλε. Και εγώ και ο κύριος Κρόιτσμαν δουλεύουμε για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει το λόγο. Μα αποσπάσει την προσοχή και τα καταφέρει θα του δώσω το λόγο. Λοιπόν, πρώτα σκιώδει εισηγητές και μετά έχω και άλλου πέντε ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, μη μακρηγορήστε για να ακούσουμε και του υπόλοιπου συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Έγγελ πρώτα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, Uh, commenting on uh, Θα ξεκινήσω σχολιάζοντας τη μέθοδο εργασίας που επέλεξε ο εισηγητής, λέγοντας ε, ότι εμείς ως ομάδα και εγώ προσωπικά ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ακολουθήσουμε την, ε, τις διαδικασίες που προτείνει και το, Συμβούλιο και για, την... Ε, για, για τις συστάδες ομάδες που πρότεινε ο εισηγητής. Ε, πιστεύω ότι οι τέσσερις βασικές συστάδες που παρουσίασε ε, νομίζω ότι θα μας δώσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με την τρέχουσα νομοθετική κατάσταση στον τομέα και πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό όμως δεν σημαίνει βέβαια ότι τα έχουμε ήδη όλα επιτύχει όσον αφορά την απλούστευση, την ασφάλεια δικαίου, την ε, ε, αποσαφήνιση. Το κείμενο ε, ναι μεν έχει στόχο να επιτύχει τους στόχους αυτούς, αλλά οι λεπτομέρειες του μπορεί να μην είναι απολύτως συμβατές με τους στόχους αυτούς και πρέπει να το επεξεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι δεν θα κάνουμε τα πράγματα πιο περίπλοκα αντί να τα απλοποιούμε. Και κυρίως για τις μικρότερες εταιρείες. Θα ήθελα της εξ αρχής να πω ένα πράγματα, γιατί μπορεί να διαχωρίζονται έτσι κάπως οι απόψεις. Υπάρχει το θέμα των ε, κατοφλίων με την πρόσβαση, σε σχέση με την πρόσβαση και την καινοτομία. Κάποια κράτη-μέλη έχουν την πρακτική να δίνουν ε, τη δυνατότητα ε, δημοσίων ε, προμηθειών σε μικρότερους διαγωνισμούς. Όμως αυτό δεν προβλέπεται στην τρέχουσα νομοθεσία. Θα ήταν όμως ενδεχομένως να δούμε τέτοιου είδους παραδείγματα που υπάρχουν στις εθνικές νομοθεσίες για να δούμε κατά πόσο έχει νόημα κάτι τέτοιο και βλέπω ότι ε, ένας δανός ε, με κοιτάει, μάλιστα δανός ε, στο γραφείο μου μου επέστησε την προσοχή σε αυτό το σημείο εχθές. Ίσως θα πρέπει να εφεύρουμε και ένα επιπλέον καθεστώς το οποίο θα μας διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αυξήσουμε κάπως και το κατώτατο όριο, το κατόφλι, ώστε πέρα από αυτό να ε, κάνουμε διαγωνισμούς που θα ε, ευνοούν τις μικρότερες ε, καινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας για το θέμα αυτό. Κάτι ακόμη το οποίο πρόσεξα και νομίζω ότι ευθύ εξ αρχή πρέπει να το θέσουμε, γιατί δεν υπάρχει επιλογή, είναι οι άμεσε πληρωμέ ε, στου ε, υπεργολάβου. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν ε, κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απλώς ένας ενδιάμεσος και, και ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας δεν θα μπορούμε να ασκήσουμε κανένα έλεγχο. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχθούμε έτσι απλά. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν με την πρόταση αυτή, αλλά νομίζω ότι οι νομικές ανησυχίες είναι πολύ ε, σοβαρότερες. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω γιατί πιστεύω ότι θα μας δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα διαδικαστικής και νομικής ε, φύσεως ε, αν το επιτρέψουμε την ε, τα θέματα της βιωσιμότητας για τις συμβάσεις των υπερκολάβων. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα πράγματα σε ένα επίπεδο ε, διαχείρισης ε, και ελέγχου που να είναι ε, δυνατόν. Γιατί αν αφήσουμε τα πράγματα στους υπεργολάβους, νομίζω ότι πράγματι αποδυναμώνουμε τις συμβάσεις και δημιουργούμε ένα καθεστώς το οποίο στο τέλος θα μας οδηγήσει σε πάρα πολλές υποθέσεις στο δικαστήριο. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Πολλά ουσιαστικά θέματα κατά την άποψή μου. Τόσοι ή άλλως έχουμε χρόνο κατά τους ερχόμενους μήνες να τα συζητήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. σε ευχαριστώ πολύ. Δίκιο έχετε που επικεντρώνεστε σε αυτά τα βασικά ζητήματα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχήν, συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Σάγκερ πιο πριν. Το χαιρετίζουμε ότι υπάρχει αυτή η πρόταση οδηγίας. Όλοι προσδοκούσαμε να την δούμε. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε μια, έναν εξυγχρονισμό χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για το 1 πέμπτο, εν πάση περιπτώσει, του ΑΕΠ. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό και για την ελεγκτική δραστηριότητα που έχουμε για τον προπολογισμό στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες αφορώνται οι χώρες αυτές για τα κονδύλια φορολογουμένων που διατίθενται σε αυτές τις διαδικασίες. και στις δημόσιες προμήθειες δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα τα επιθυμούσαμε και δεν υπάρχουν τόσο σαφείς κανόνες. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τώρα ότι υπάρχουν εδώ σαφείς κανόνες τον κύριο Ταραμπέλα θέλω να τον ευχαριστήσω για το έγγραφο εργασίας που δίνει μια πολύ καλή επισκόπηση σε ομάδες και κατηγοριοποίηση των θεμάτων. Είναι πολύ καλό να δουλεύουμε με clusters, με κατηγορίες και ομάδες. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Στην ομάδα 2, cluster 2, συμμερίζομαι την άποψη του Φρανκ Έγκερ ότι όσον αφορά τις υπεργολαβίες υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν, να υπάρξουν προβλήματα και με τις άμεσες πληρωμές υπάρχει άμεσο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όπως το διατύπωσε ο ε, κύριος Έγκερ, δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, να γίνονται τέτοιες ε, άμεσες πληρωμές σε υπεργολάβους. Και εγώ το θεωρώ, με τον ίδιο τρόπο το βλέπω, διότι θα άλλαζε το πλαίσιο των πραγμάτων εκβάθρων σε πολύ σημαντικό βαθμό. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν και πολύ δύσκολα πράγματα. Τα κοινωνικά κριτήρια, ο κύριο Ταραμπέλα δίνει μεγάλη αξία σε αυτά. Καλώς ε, βαίνει καλώς αυτό, εντάξει με τα κοινωνικά κριτήρια, αλλά να μην είμαστε τόσο υπερβολικοί και μειώσουμε τη συμβατική ελευθερία των συμβαλόμενων. Αυτό θα μπορούσε να είναι δύσκολο για να μα βοηθήσει να πετύχουμε τον άλλο κύριο στόχο, δηλαδή υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι άμεσε πληρωμέ βρίσκονται στην κατηγορία Cluster 5 και η όλη κατηγοριοποίηση σε, σε αυτές τις ομάδες, σε δύο ας το πω έτσι στρατόπεδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες. Το κατόφλι θα μπορούσε να το παρακάμψει κανείς. Πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε οι στόχοι μας. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούστηκε. Ναι, αλλά πρέπει να προσέξουμε και τους άλλους στόχους που έχουμε να μην αντιφάσκουμε με αυτούς. Να ασχοληθώ τώρα με την υποκατηγορία «Cluster 10 Πρόκειται για ορισμούς ορολογίας, για το scope, το εύρος, το φάσμα. Πρέπει να προσέξουμε να μην εμπλακούμε στις αρμοδιότητες άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Ευρωκοινοβούλιο και για αρμοδιότητες που δεν έχουμε να μην δράσουμε επί θεμάτων που δεν έχουμε αρμοδιότητες και από πλευράς Επιτρόπου γνωρίζω ότι υπάρχει ε, προσπάθεια που γίνεται αλλά για την στεγανοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση που θα δημιουργεί σύγχυση. Πρέπει σε κάποιους ορισμούς να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αν θέλουμε να είμαστε σαφείς πρέπει και οι ορισμοί να είναι σαφείς. Τι είναι σύγκρουση αρμοδιοτήτων και συμφερόντων. Δεν είναι σαφές. Τι είναι οι προνομιακές σχέσεις, links, δεν είναι σαφές. Τι σημαίνει ενδεδειγμένο, κατάλληλο, appropriate. Δεν είναι και αυτό σαφές. Και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα σταθμίσουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα, το κριτήριο χαμηλή τιμή είναι το ίδιο ή διαφορετικό σε σχέση με το βάρος του, με το οικονομικό προτέρημα. Δεν νομίζω λοιπόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα για τις προσφορές, τις χαμηλότερες οικονομικές προσφορές. meet. Ε, και πρέπει να έχουμε έναν ανεξάρτητο φορέα που θα υποπτεύει δημόσια τα πράγματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γραφειοκρατική επιβάρυνση. Απλώς το επισημένο ευχαριστώ. Η κυρία Ρούιλε, σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη σαφή δομή με αυτή τη σαφή δομή μπορούμε να δουλέψουμε καλά και αποτελεσματικά. Θέλω να διασφαλίσω ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον θα προσπαθήσω να προχωρήσουμε έτσι. Για που ω μικρότερη ομάδα θα έχουμε ίσω απλούστερο έργο απότερου. Όμω ε, ο συντονισμό και με τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ πρέπει να διασφαλιστεί και στην ίδια την κοινοβουλευτική μα ομάδα και στι άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Να μην υπάρχουν ασυντόνιστε, μη συμπεφωνημένε τροπολογίε και δημιουργηθεί σύγχυση. Θα κάνω προσπάθεια να πετύχουμε αυτό το στόχο. Όμω κάπω έχω και εγώ κάποια προβλήματα με τα κέντρα βάρος που θέτεται και πρόσεξα ότι κάποιοι συνάδελφοι άλλα σημεία προανέφεραν. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ξεκινήσω με την ομάδα Cluster 10 για το φάσμα, το εύρος εφαρμογής, διότι το πεδίο εφαρμογής είναι ένα κύριο σημείο από το οποίο άλλα πράγματα μετά ρυθμίζονται εφ' εξής. Θα λυπόμουν αν δεν βρισκόταν αυτό στο επίκεντρο. Επίσης το θέμα της ε, δημόσιας ε, συνεργασίας ε, και υπό τον ορισμό στο άρθρο 1 υπό το φάσμα, εδώ θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλω να επισημάνω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί άμεσα. Λέτε ότι πρέπει ε, περιορισμένη συμμετοχή ιδιωτών να προβλέπεται σε τέτοιες ε, δημόσιες ιδιωτικές συνεργασίες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει διάφορες αποφάσεις που έλαβε. Κρούω κόδωνα κινδύνου να μην εντάξουμε πράγματα εδώ που δημιουργούν νομική αβεβαιότητα και ανασφάλεια που θα δημιουργήσουν μετά ανάγκη πολλών προσφυγών στο 10. Διότι εδώ είναι δύσκολο το πράγμα του διαχωρισμού δημόσιας ιδιωτικής σύμπραξης. Πρέπει να είναι σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές. Όταν πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα πρέπει να έχει, υπάρχουν, να έχει προτερήματα έναντι άλλων συμπράξεων. Αυτό το οποίο είναι σωστό είναι το ότι αναφέρεται το θέμα των συνεταιρισμών και τη συμμετοχή συνεταιρισμών εδώ υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα στη συμμετοχή συνεταιρισμών. Πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτά τα προβλήματα που μέχρι στιγμής δεν βρίσκονται αυτές οι λύσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να αναφέρω και την ομάδα κατηγορία κλάστερ 9. Και εγώ έχω προβλήματα με αυτό το φορέα, ε, φορέα ή θεσμό απελευθέρωσης. Γιατί χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στο δημόσιο κεντρικό τομέα. Και εδώ πρέπει να διαρωτηθούμε για την αναλογικότητα των μέσων και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα θέματα. Διότι εδώ αφορώνται θέματα δήμων και κοινοτήτων και πρέπει να γίνουν δεκτά αυτά και υπάρχουν ήδη δομέ και διαρωτώ τι θα κάνει μια τέτοια ρυθμιστική αρχή. Έχουμε και νομικές δομές ε, με την οδηγία για τα νομικά μέσα. Λοιπόν, δεν βλέπω καθόλου να υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αυτή η αρχή, η ρυθμιστική αρχή όπως προτείνεται. Για τα άλλα σημεία τώρα. Και εγώ κάπως προβληματίστηκα με το σημείο 2, κλάστερ 2, κατηγορία 2 δια... ανεφεί το ερώτημα για μένα γιατί δεν υπάρχει εδώ διασύνδεση με τον εντολέα ή την ε, παραγγελία. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει, κατεπηγόντως. Όταν περνάμε στις δημόσιες συμβάσεις, ε, τότε πρέπει να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά το δεσμό του εντολέα ή της παραγγελίας. Ε, διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να αρχίσουν κάποιοι να, να αναφέρονται σε θέματα διαφθοράς ή εσχροκέρδειας. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και σε σχέση με το υπιότερο καθεστώς το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα, Τώρα αποδυναμώνεται αυτό και μόνο για πολύ λίγες υπηρεσίες ε, μπορεί να εξετάζεται. Υπενθυμίζω όμως την γνωμοδότησή μας για τη διασφάλιση των ε, υπηρεσιών Α και Β κατηγοριών. Δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να διαλυθούν αυτές ή να αποδυναμωθούν και για το θέμα της ε, κατηγορίας 4. E-procurement, ε, ηλεκτρονικές προμήθειες. Ε, το πρόβλημα, το ερώτημα είναι για την διετή περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 είχε προβλέψει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τις ηλεκτρονικές αυτές συναλλαγές. Από 15% 5% τώρα έχουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι καταλήξαμε σε μια διετία, σε μια κατάσταση όπου η υποχρεωτική εισαγωγή ηλεκτρονικών τέτοιων προμηθειών ε, διασφαλίζεται. Πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη και για την ανάπτυξη αντίστοιχων δομών και διαρθρώσεων που πρέπει να είναι δεδομένες για να προχωρήσουμε και η συμβατότητα των, πλα, των ε, πλατφορμών ε, των ε, δυνατοτήτων δράσεων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Now I'm going to be sharing Θα δώσω το λόγο στον κύριο και παρά το γεγονός ότι είμαι και εγώ το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, μια μικρή ομάδα σαν τη δική μας ε, μοιραστήκαμε τα καθήκοντα γιατί έχουμε ένα ε, μεγαλύτερο και ένα νεότερο συνάδελφο και έτσι τα μοιράσαμε τα καθήκοντα. Το θέμα των δημοσίων προμηθειών αφορά όλες τις δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εμείς επικροτούμε την πρόταση της Δανικής Προεδρίας και συμφωνούμε και με την κατηγοριοποίηση στις 10 αυτές ομάδες. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι περισσότεροι από τους συναδέλφους. Μόνο απλώς ε, να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου ε, σε σχέση με την ε, υπερνομοθέτηση, την υπερρύθμιση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο, πολύ επιπλέον άχθος. Πρέπει να επιτρέπει στην, στην αγορά να λειτουργεί εύρυθμα. Ναι, λέει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ζητήματα γύρω από τη στρατηγική χρήση ε, των προμηθειών να μην είναι τόσο ε, ρυθμισμένα ώστε να καταστρέφουν οποιαδήποτε ασφάλεια δικαίου ε, και να μην δημιουργούν προβλήματα στο, στην πιο συμφέρουσα προσφορά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό ως εναλλακτική επιλογή αλλά όχι ως εναλλακτική επιλογή και ε, αντικατάσταση αυτών που θα έπρεπε οι δημόσιες αρχές να κάνουν εκείνες. Ίσως ε, δεν ε, νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε το ρόλο των δημοσίων αρχών ε, σε σχέση, για παράδειγμα, με την ε, άτυπη, παράτυπη εργασία ε, στον δημόσιο τομέα. Ό,τι λοιπόν πρέπει να γίνει από τις δημόσιες αρχές πρέπει να γίνεται από αυτές. Και πιστεύω ότι κάποιες από τις ιδέες μας πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ επιλεκτικοί. Το στρατηγικό αυτό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια φαντάζομαι ότι θα δεν θα σας εκπλήξω όταν σας πω ότι το νέο μέσο για τις ε, καινοτόμες ε, ε, δημόσιες συμβάσεις είναι τη, τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που θα κάνουμε με τον κύριο Κόσνικ είναι να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο. κύριος Διόν και μετά ε, ο κύριος Ζουβέν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ταραμπέλα για αυτό το έγγραφο εργασία. Η μέθοδο που υιοθέτησε είναι σωστή και η κατεύθυνση στην οποία στοχεύει το έγγραφο σωστή και μα χαροποιεί ω κοινοβουλευτική ομάδα. Για μα είναι μια εξαιρετική βάση για τη δουλειά μας. Τώρα, κάποια σημεία. Κλάστερ 1. Γνωρίζω βάσει πείρας με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές μας ότι ακριβώς αυτή η διαδικασία όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε ολόθερμα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό και διευκολύνει τα πράγματα. Αυτές οι νέες εγγυήσεις. Οι νέες εγγυήσεις δεν θα πρέπει να είναι γραφειοκρατικού χαρακτήρα, να μην δημιουργούν γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αυτή η διαδικασία ήταν πολύ καλή. Ομάδα Cluster 2 σε αντίθεση με άλλους προλαλήσαντες χαιρετίζω, εγώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ξεχωριστά κοινωνικοί στόχοι θα λαμβάνονται υπόψη. Εδώ θα ήθελα όμως τους μισθούς ε, να το, να τα έχουμε ως ε, σημεία. Δεν συμφωνώ με τον κύριο ε, Προλαλήσαντα ότι υπερβαρύνονται ε, με αυτές τις προτάσεις τα πλαίσια. Είναι πτυχές που επανειλημμένα στις δημόσιες συμβάσεις και τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, διότι Όσοι υποβάλλουν προσφορές διαρκώς προσπαθούν να κάνουν κοινωνικό dumping ώστε να πάρουν την παραγγελία και τη σύμβαση, τις δημόσιες αυτές συμβάσεις. Πέρα από αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις σε όλες τις πτυχές. Η υπεργολαβία φυσικά είναι ένα πρόβλημα. Αν όμως με κάποιον που υποβάλλει προσφορά υπάρχει μια συμφωνία που όμως προβλέπει μετά στη συνέχεια υπεργολαβία και μικρότερη προσφορά, ε, τότε κάποιος άλλος ε, θα είναι ο ε, υπεύθυνο και αυτό δεν είναι καλό. Τώρα για τις προδιαγραφές και στο κοινωνικό επίπεδο και στην Ολλανδία εδώ έχουμε έντονη συζήτηση που διεξάγεται. Στην πρακτική εφαρμογή τι γίνεται, δεν γίνεται δεκτή η πρόταση αυτή που να λέει ότι για παράδειγμα τα μανιτάρια θα πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να καλλιεργούνται, αλλά θα πρέπει πάντα οι εργαζόμενοι να την χάνουν σωστή αντιμετώπιση. Για τέτοιου είδου ετικέτε λοιπόν ε, στα μανιτάρια από τους παραγωγούς πολλές φορές δεν γίνονται δεκτέ αυτές οι προτάσεις. Πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα σε όλε του τι πτυχέ. Για τι άλλε προτάσει κλάστε ομαδοποιημένε, συμφωνώ είναι πολύ ε, καλές και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις, στους χρονικούς περιορισμούς ε, ως διορίες. Οι ε, παραγωγοί μου το επισήμαναν. Όταν είναι πιο στενές οι προθεσμίες, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούνται δυσκολίες. Και συμφωνώ και με την κατηγορία Cluster 9. Εδώ άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν επιφυλάξεις τι θα Πώς θα πρέπει εδώ η εποπτεία και οι δράσεις να διοργανωθούν. Είμαστε, ας το πω υπάρχει μια κόποση όσον αφορά φορείς, υπηρεσίες και θεσμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς αποκλειστικά να μπορούμε εμείς όλα να τα προβλέπουμε. Επίσης όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη συνεργασία. Συνεργασία με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Αυτό το επιθυμούν να, έχουν, να το έχουν ως δυνατότητα πολλές τοπικές αρχές. Στην πρακτική εφαρμογή δυσκολεύονται όμως τα πράγματα. Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Γι' αυτό χαιρετίζω το γεγονός ότι ο εισηγητής ανάφερε αυτό το θέμα. Θα δώσουμε λοιπόν ε, έτσι με αυτόν τον τρόπο στον πρώτο γύρο σε εσάς της παρεμβάσης σας. Συνάδελφοι πρέπει να πω ότι έχουμε μια στιγμή πόσους εννέα αγορητές που ζητούν να παρέμβουν. Θα ήθελα να έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο χρόνο και δεν θέλω να δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τον κύριο Ζουβέν. Καθένα δύο λεπτά το μέγιστο για τι παρεμβάσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σα πω ποιοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο. Αν κάποιοι θέλουν να. Mr. Baldessari, Mr. Arias, Mr. Mr. Mr. Schwab, Mrs. Mr. Obermeyer. Σα διάβασα τα ονόματα για να αφαιρέσει κάποιο την παρέμβασή του αν Δύο λεπτά ο καθένα λοιπόν. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά θα υπάρχει και ευκαιρία στη συνέχεια να υπάρξει η παρέμβαση. Ξεκινάμε με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή την οποία εξέθεσε ο εισηγητή μα σήμερα το πρωί για την απλούστευση των κανόνων και ρυθμίσεων και να υπάρχει η διασφάλιση αρκετή ευελιξία με ε, αφαίρεση με διαγραφή τη νομική αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Καθώ υιοθετήσαμε αυτή τη γραμμή στην αρχική μα έκθεση και όσον αφορά την πιο συμφέρουσα προσφορά, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα, που πολύ σωστά ο Μάρκο Ταραμπέλα ανέφερε, είναι να είμαστε σαφέστεροι στους ορισμούς. Η σαφήνεια στους ορισμούς νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των τροφικών, των τροφίμων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα τι σημαίνει τοπικά παραγόμενο προϊόν τι γίνεται εδώ σε σχέση με τα διασυνοριακά μεθοριακά, πώς θα δώσουμε ίσο, ισοδίκαιο πεδίο για όλους τους παραγωγούς και τους μικρούς ε, και μικρομεσαίους παραγωγούς σεβόμενοι πάντα την επιθυμία να μπορούν με τοπικά προϊόντα να τρέφονται και να καλύπτουν τις ανάγκες τους οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και εδώ πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Το άλλο είναι οι δημόσιες συμβάσεις για τους αποκαλούμενους παθητικούς καταναλωτές στα νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία και αλλού όπου σητίζονται. Έχουν το ίδιο δικαίωμα να διασφαλίζεται αναβαθμισμένη υψηλή ποιότητα στα προϊόντα που καταναλώνουν και να μην έχουν μόνο τα πιο φθηνά προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα για αυτούς. Ένας τους τρόπου για να διευκολύνουμε την πρόσβαση είναι σε σχέση με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, το ότι θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και ευφυεί όσον αφορά τον διαχωρισμό των ε, προμηθειών σε κατηγορίες και πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα να καλύπτονται έτσι οι ανάγκες. Τα κοινωνικά κριτήρια, συμμερίζομαι την άποψη, δεν πρέπει όλα να τα συγχαίουμε εδώ. Ελευθερία συμβατική συνάψης συμβάσεων και αυτό είναι σημαντικό. Πώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε ή να ετικετοποιήσουμε οι κανονισμοί, οι κανόνες ε, για αυτά τα προϊόντα είναι εθνικοί και φυσικά πρέπει να είναι σεβαστοί. Αλλά δεν νομίζω ότι για την νομοθεσία για προμήθειες πρέπει να επιβαρύνουμε με πρόσθετους κανονισμούς που ισχύουν για τα κράτη μας. Και ένα θέμα προς τον κύριο Ταραμπέλα για το θέμα των ευάλωτων ομάδων, εξαιρέσεις για ευάλωτες ομάδες την ε, προσθήκη για το προσιτό των τιμών και το, προσπελάσιμο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων ατόνων με αυτά τα προϊόντα. Ο κύριος Μπαλτασάρη, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ ζητώ τον κύριο Ταραμπέρα, τον οποίο ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανε, να κάνει μεγαλύτερη εμβάθυνση ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται με τη διαδικασία όσον αφορά το, να, τι γίνεται με τη χαμηλότερη, την πιο υποφελή προσφορά την οικονομικά. Η διαδικασία όσον αφορά τη χαμηλότερη τιμή είναι μεγάλο πρόβλημα κυρίως για δημόσια έργα. Ε, συστηματικά η δημόσια διοίκηση προωθείται να χρησιμοποιεί αυτή την ε, προσέγγιση διότι αποφεύγει την παρέμβαση άλλων λεκτικών φορών ε, στη χώρα μας πάνω από 50% είναι οι αναθέσεις που γιονται την χαμηλότερη τιμή. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια για περιβάλλον, για ποιότητα, κοινωνικές πτυχές. Όταν οι επιχειρήσεις για να βρουν δουλειά σε μια στιγμή κρίσης όπως είναι αυτή δέχονται μείωση τη τάξη 40, 50, 55%. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα πρέπει να διορθωθεί και θα πρέπει να βαθυθεί η ανάλυση. Άλλη πτυχή, ε, σε μια πολύ συνολική ρύθμιση που θα πρέπει να κατευθύνεται κατά τομέας. Οι αναθέσεις ε, ε, για τις οικοδομές είναι διαφορετικές από άλλες αναθέσεις. Γενικά κριτήρια που ισχύουν για όλους είναι κάτι δύσκολο. Αλλά το, επι, το επιβάλλει η γενίκευση. Όμως κάποια κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να θεσπιστούν και σε αυτή την οδηγία κυρίως ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε στους επιχειρηματίες μας ε, όσον αφορά τον αγωνισμό ε, να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι των, ε, των εταιριών από το εξωτερικό. Ε, να παρέχουν και αυτές που, που συμμετέχουν οι εταιρείε του εξωτερικού να, να πρέπει να πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτασάρη. Μιλήσατε εντός διλεπτού και ο κύριος Αρίας είναι ο επόμενος θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανε ο κύριος Ταραμπέλα. Είναι μια καλή αρχή ως αφετηρία. Εγώ μια και έχω δύο λεπτά θα πρέπει να αναφερθώ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πτυχές αυτές. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να ανοίξουμε την πόρτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο τέλος τέλος είναι εκείνες που υποστηρίζουν και διατηρούν την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι λοιπόν ένα καλό εργαλείο, ένα καλό μέσο το ηλεκτρονικό εμπόριο για να γίνεται αυτό. Η διαφάνεια έχει θεμελιώδη χαρακτήρα και νομίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο το ηλεκτρονικό εμπόριο και στις ε, προμήθειες αυτές ηλεκτρονικά για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ας το πω έτσι, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τον εποτισμό και να υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουν οι πύλες, ε, οι θύρες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους να συμμετέχουν σε αυτές τις διαργασίες όπως οι μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις. Για τις πιο φθηνές τιμές στις προσφορές ε, και εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Η δυνατότητα να γίνουν όλα αυτά πιο διαφανή και η απλούστευση είναι σημαντικές υποθέσεις. Να ανοίξουμε τις πόρτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να διευκολύνουμε διευκολύνουμε να έχουμε καλύτερες προσφορές και τιμές όσον αφορά τις δημόσιες αυτές συμβάσεις. Για τα θέματα των δεδομένων και με μια τέτοια οδηγία η προστασία δεδομένων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα πρέπει να συζητήσουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με αυτό. Και τέλος τέλος πιστεύω ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή και είναι θεμελιώδης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Είναι σημαντικά θέματα η διαφάνεια και η απλούστευση και νομίζω ότι για αυτού του είδους τις συμβάσεις θα έχουμε μεγάλες ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Uh, very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Κοφεράτη και Σαρντεμόζε. Και Κοφεράτη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, έκανε έξοχη δουλειά ο Μάρκ και συμφωνώ πάρα πολύ με το αίτημα που έκανε να ε, τη συνέχεια των συζητήσεων να, και στην, να, να το στέσουμε και στις πολιτικές ομάδες. Οι δημόσιες προμήθειες είναι σημαντικός μοχλός για την ε, ανάπτυξη θα πρέπει να προστάσουμε σε κάποια συμπεράσματα γρήγορα προς όφελος όλων των χωρών, αλλά είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και ο κίνδυνος είναι να υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των απόψεων διαφόρων επιτροπών και τελικά να υπάρχει μια διάχυση πολύ μεγάλη των ιδεών και χρονικά. Είναι σημαντική η αναβολή, αν θέλετε, να βρούμε έναν τόπο. Η πολιτική ομάδα είναι ιδεώδης χώρος, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τις διάφορες απόψεις που θα επικρατούν. Όσον αφορά μετά πιο συγκεκριμένα την ουσία, ε, πιστεύω πάρα πολύ στην αποτελεσματικότητα της ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες. Η ευελιξία είναι ένα πράγμα. Αν η ευελιξία όμως μεταμορφωθεί σε τόσες υποθέσεις διαφορετικής πρόσβασης, κινδυνεύουμε να ανοίξουμε το χώρο σε λανθασμένη διαχείριση και επικίνδυνη ε, όσον αφορά την ανάθεση. Τώρα όσον αφορά την ομάδα 2, το cluster 2, συμφωνώ με αυτά, με τις παρατηρήσεις που άκουσα. Η μέγιστη μείωση των τιμών, η χαμηλότερη τιμή είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αδιαφάνεια και στην έλλειψη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που δεν είναι μόνο αυτά των ατόμων που συμμετέχουν. Μετά, η πιο υποφελής οικονομική προσφορά αγκιάται την ποιότητα και μια επαλήθευση πιο συνολική από πλευράς ε, των φορέων που ενεργοποιούν την όλο διαγωνισμό προσφορά και όχι τιμή. Προσφορά πιο οικονομική, πιο υποφελής οικονομικά και όχι χαμηλότερη τιμή. Μετά στον αφενταξινόμηση. Πιστεύω ότι ο μόνο ε, τομέα, σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε και για την ομοιομορφία που χρειάζεται διάκριση με τι διαδικασίες, είναι οι κοινωνικέ υπηρεσίε. Οι άλλοι τομεί λίγο πολύ είναι παρεμφερεί, παρόμοια. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαλτεμόζε. Και μετά ο κύριος Φαμπ. Κυρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η απλοποίηση είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πρότασης αυτής και εμείς τον υποστηρίζουμε. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Οπότε θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Έγγελ να λάβουμε υπόψη ένα καθεστώς ε, κάπως πιο ελαφρύ, να αυξήσουμε το κατόβλι και να έχουμε ένα καθεστώ δημοσίων συμβάσεων για ένα χαμηλότερο κατόφλι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπω πιο ελαφρύ, με λιγότερου κανόνε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Το έχουμε στη Δανία. Ξέρω ότι το έχουν και άλλε χώρε. Και επίση ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα συμφωνούσε με μια τέτοια προσέγγιση. Ε, επίση, θα δίναμε καλύτερε ευκαιρίε ε, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμμετέχουν γιατί η γραφειοκρατία ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο δύσκολο για τις κυβερνήσεις, αλλά είναι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ένα πιο ελαφρύ καθεστώς με λιγότερους κανόνες, όπως επίσης και να αυξήσει το κατόφλι. Η κυρία Ρούλε κάτι είπε εκτός μικροφώνου που δεν ακούσαμε. καλά κάνει ο εισηγητής ε, που υποστηρίζει το κατόφλι το υπάρχον. Απλώς πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, πρόεδρος, νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία, ιδανική προεδρία με τη δική σας υποστήριξη να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη Δανία. Ο κύριος Ταραμπέλα θα το λάβει υπόψη. Σφαμπ, Γκέπχαρτ και Καλνιέτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα. Πρώτον για το θέμα των αποκαλούμενων εθνικών ε, φορέων. Δεν προτείνεται αυτό από την Επιτροπή για να υπάρξει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, αλλά για να έχουμε καλύτερη εποπτεία των ε, εξελίξεων στα κράτη-μέλη και του τι συμβαίνει εκεί μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε όσον αφορά τις, ε, την οδηγία για τις ε, ε, άδειες αυτές. Μία από τις, ε, ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι μόνο τότε έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα στοιχεία όταν γίνεται κάποια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει νέα γραφειοκρατική επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά όμως η σκέψη για την ενιαία εσωτερική αγορά στην εξέταση των αριθμών και αριθμητικών μεγεθών να βρει τη σωστή θέση. Δεύτερον, για τον τον διάλογο και την, ε, ε, όπου το αναφέρει ο κύριος Ταραβέλα στο έγγραφο συζήτησης ως σημαντικό στοιχείο. Ναι, αλλά υπάρχει γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που λέει να μην υιοθετηθεί μια διαφορετική διαδικασία από ότι οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις και οι προσφορές για την σύναψη συμβάσεων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να προταθεί να γίνει αυτό. Μπορεί και στο μέλλον να ενισχύεται η συνθήκη αυτή. Καταρχήν δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα. Για την αμοιβαιότητα μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτά που είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης. Για το θέμα όσον αφορά την ίδια την σύναψη, συμφωνώ με την κυρία Ρούλε. Και για το value for money δεν θέλω να αναφερθώ σε θέματα τα οποία αναφέρθηκαν πιο πριν από την κυρία Κοράτσα Μπίλντ, Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα κατά της αηφορίας και των κοινωνικών κριτηρίων. Αλλά αυτά τα κριτήρια πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αμερόληπτα ουδέτερα στην εφαρμογή τους. Δεν θέλουμε να υπάρξει κατακαιρματισμός, κατάτμιση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτά που στο πέμπτο σημείο νομίζω αναφέρει ο κ. Ταραμπέλα, ότι χρειάζονται τικέτες που θα αντανακλούν μια αξιοπιστία. Εδώ είναι το αποφασιστικό στοιχείο και ε, δεν είδαμε να υπάρχουν κάποιες ε, προτάσεις σχετικά. Αναμένουμε να δούμε τι θα προταθεί στη συζήτηση. Περνάω στο τελευταίο ηλεκτρονικές συμβάσεις. Μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο όταν τα εθνικά συστήματα μπορούμε να τα συνδέσουμε μεταξύ τους καλύτερα. Έτσι νομίζω μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Η κυρία Γκέπα τώρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μια πολύ καλή προσέγγιση του Μαρκ Ταραμπέλα για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων και τις φοβίες που υπήρχαν, οι δισταγμούς το ότι θα ήταν μια δυσχερέστατη ακαθόδη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο αυτά δείχνουν, καταδείχθηκε ότι είναι αβάσιμα και αυτό είναι σημαντικό. Σε δύο σημεία θα επικεντρωθώ σήμερα. Το πρώτο από αυτά είναι το θέμα των πιο φθηνών προσφορών των φθηνότερων προσφορών και στην τελευταία αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τις συμβάσεις ε, το είχαμε συζητήσει και βρήκαμε μια καλή βάση εργασίας με το Συμβούλιο. Είπαμε δεν είναι το σημαντικότερο η φθηνότερη προσφορά αλλά η πιο ευνοϊκή προσφορά. Η πιο ευνοϊκή προσφορά σημαίνει η ποιότητα των προϊόντων να λαμβάνεται υπόψη αλλά να λαμβάνονται επίσης υπόψη και κριτήρια που αφορούν την αηφορία όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη στην οποία θα θεμελιώνουν αυτή την προσέγγιση που τότε στο παρελθόν υιοθετήσαμε δεν πρέπει πάλι να την εγκαταλείψουμε και είχα την εντύπωση σήμερα στη μία ή άλλη παρέμβαση συναδέφων ότι θα μπορούσαμε εκεί να καταλήγαμε. να κινδύνου, να μην το κάνουμε αυτό. Να είμαστε επακριβέστεροι, πιο εξειδικευμένοι, πώ βλέπουμε και θέλουμε να καλύπτονται αυτά τα κριτήρια. Με αυτό θα συμφωνούσα. Αυτό σημαίνει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε με κανένα τρόπο αυτέ τι αρχέ. Το δεύτερο θέμα, και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, και στην έκθεση τη κυρία Ρούιλε το είχαμε συμπεριλάβει έτσι, και στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία είχε εγκριθεί είναι το θέμα των υπεργολαβιών, των υπεργολάβων που θέλουμε τώρα να το αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο. διότι σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα στις οικοδομές, με μεγάλες τέτοιες ε, συμβάσεις, ήθιστε μια εταιρεία να αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός έργου, αλλά η δουλειά να γίνεται από υπεργολάβους. Ε, τότε δεν ωφελεί τίποτα αν έχουμε την κύρια επιχείρηση που απαιτούμε από αυτήν να σέβεται αυτά τα κριτήρια, αλλά οι υπεργολάβοι δεν τα σέβονται στη συνέχεια. Έτσι παρακάμπτονται τα πράγματα και θέλουμε πολιτικά να αποφύγουμε την παράκαμψη αυτή. Και αυτό αφορά και την ποιότητα. Και φυσικά έχουμε και το θέμα που πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη, το ότι σήμερα πολύ συχνά βλέπουμε σε μεγάλες τέτοιες συμβάσεις και παραγγελίες ότι οι τιμές που ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με 10, 20, 30% υπάρχει απόκληση. Η τελική τιμή είναι πολύ υψηλότερη στο τέλος τέλος και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη συζητήσεις. Ευχαριστώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, αυτό είναι και το θέμα προς διαπραγμάτευση. Κυρία Κανιέτη και ο κύριος Όμπερμαϊρ. Κυρία Κανιέτη πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρκ Ταραμπέλα, τον εισηγητή, για τις ε, προτάσεις του. Θεωρώ ότι οι σημαντικότερες αρχές είναι η απλούστευση και η διαφάνεια. Και σε αυτό το πνεύμα πιστεύω ότι η χρήση της διαδικασίας που είναι ανταγωνιστική με διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επεκταθεί και να γίνει μια τυποποιημένη διαδικασία που θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Εξίσου σημαντικό όσον αφορά τα κριτήρια είναι η εξάλληψη του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής και μόνο δεν είναι κάτι που πάντα δικαιολογείται ως κριτήριο, γι' αυτό θα πρέπει να επεκτείνουμε την πλέον εποφελή οικονομικά πρόταση ε, για όλες τις διαδικασίες. Όχι μόνο για τις συμπράξεις για την καινοτομία και τον ανταγωνιστικό διάλογο, όπως προτείνεται. Κλείνοντας, πιστεύω ότι όχι μόνο οι, ανα, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν οικονομικούς φορείς που παραβιάζουν υποχρεώσεις όσον αφορά φόρους, κοινωνικό, περιβαλλοντικό νόμο και δείχνουν συνεχείς ελλείψεις σε πρώτερες επιδόσεις, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν δεσμευτικές προδιαγραφές για τον αποκλεισμό τέτοιων εμπορευομένων. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ που δώσατε τόσο κομψό παράδειγμα. Ο κ. Σόμπερμαια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ και εγώ. Σημείο πρώτο. Η σημασία που θα πρέπει να αφήνουμε περιθώρια για τις τοπικές αρχές και την αυτοδιοίκηση σε θέματα της ε, ευημερίας, κοινωνικής ευημερίας. Πολύ σημαντικό και με δύο παραδείγματα να καταδείξω ότι ενώ δεν είμαι ευτυχής για το ότι τα κριτήρια αυτά για τέτοιο είδους υπηρεσίες θα πρέπει να ισχύουν. Παράδειγμα, για τις ε, υπηρεσίες διάσωσης ε, όταν έχουμε μεταφορά ασθενών και όταν έχουμε θέματα ανταγωνισμού και θέματα συμβάσεων δεν μπορούν υπό αυτό το πρίσμα να ρυθμίζονται. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η υπηρεσία της διάσωσης και μεταφοράς ασθενών που αφορά κοινωνικές προδιαγραφές, υγειονομικές προδιαγραφές και προδιαγραφές υγείας δεν είναι θέμα ανταγωνισμού και ούτε είναι θέμα το οποίο διαφορετικά μπορεί να ρυθμίζεται και φοβούμε ότι αν εδώ εντάξουμε αυτά τα θέματα στον ανταγωνισμό θα υποβαθμιστεί η ποιότητα και θα έχουμε αρνητική εξέλιξη στην μείωση των μισθών προς τα κάτω με, ως μια σπυροειδή εξέλιξη για να αναφέρω πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην καταλήξουμε σε υπονόμευση των κοινωνικών δομών των περιφερειακών και τοπικών αρχών και ε, αρμοδίων. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Ομπερμάιερ. Δώσατε πολύ καλό παράδειγμα, υπήρξατε σαφέστατος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους πάρα πολύ. Λυπάμαι, λυπάμαι που σας πίεσα χρονικά, αλλά ήταν πολύτιμες συνεισφορές και θα ήθελα να δώσω λόγο και χρόνο και στον κύριο Ζουβέν. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε ακριβώς την ώρα μας. Θα ζητήσω από τον Κλάους Βίτνερ να προβεί σε κάποια σχόλια. Αν μπορείτε σε ένα τετράλεπτο να κάνετε κάτι, θα βοηθούσε. Θα ήθελα να μιλήσει και ο συγγητή για να ολοκληρώσει και να θέσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα θέλει ο συγγητή να το κάνω εγώ. Ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινούμε το χρονόμετρο για να βλέπετε πόσο καλά τα πάτε από πλευρά χρονική. Καλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να είμαι γρήγορο και σύντομο. Να μπω στα βασικά θέματα. Πρώτο θέμα είναι το θέμα των κατοφλίων Μιλάμε για 18%-19% του ΑΕΠ του εσωτερικού. Αυτό δεν αληθεύει. Αυτό που καλύπτουν την οδηγία είναι μόνο περίπου 4 με 5%. Το να αυξήσουμε περαιτέρω το κατόφλιο θα καλύψουμε ακόμα λιγότερο μέσω των οδηγιών και θα πετύχουμε την ισότιμη βάση που θέλουμε. Διεθνέ δίκαιο, όλα αυτά, όλε τι πτυχέ θέλαμε να καλύψουμε, έτσι καλύπτουμε παρκώ ηλεκτρονικές κρατικές προμήθειες. Η Πορτογαλία μπόρεσε να το πετύχει αυτό σε 1,5 χρόνο. Άρα δεν και εμείς δεν προτείνουμε 1,5, έχουμε 4,5 χρόνια μπροστά μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περίπου 99% πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχουμε σταδιακή προσέγγιση, σταδιακή εφαρμογή. Μπορεί κανείς να είναι λοιπόν φιλόδοξος και να επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ούτε για τις αρχές ούτε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικά κριτήρια. Προφανώς προσπαθήσαμε, όπως είδατε στην πρόταση, να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε κοινωνικά κριτήρια, διατηρώντας τη διασύνδεση με το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε την ισότιμη αντιμετώπιση και ότι βρίσκουμε καλές εφαρμόσιμες λύσεις και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να βρούμε τέτοιες λύσεις αν παραστεί αναγκαίο. Το θέμα είναι της ανάθεσης μετά και τα κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια ανάθεσης θέλουμε κριτήρια που να είναι πιο οικονομικές, για πιο οικονομικές προτάσεις ε, και πιο οικονομικά υποφελείς προτάσεις, αλλά δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τις τιμές αποκλειστικά. Μπορεί να έχουμε και τυποποιημένα προϊόντα που θέλουμε να κινηθούμε μόνο βάσει ε, της τιμής και όχι βάσει κύκλου ζωής και πιο γενικά κριτήρια. Όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, έχουμε σαφή νομολογία του δικαστηρίου. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά πρόβλημα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και κάποια στοιχεία της νομολογίας φαίνεται να βασίζονται σε συνθήκη και όχι μόνο σε οδηγίες. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε αυτό και ε, όσον αφορά το να αλλάξουμε το θέμα αυτό διακυβέρνηση, εποπτική φορείς. Τι προτείνουμε, όχι να δημιουργήσουμε τεράστιες δομές και να δημιουργήσουμε προβλήματα και αύξηση της γραφειοκρατίας. Όπως είπατε, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και τα κράτη-μέλη δεν έχουν αρκετές πληροφορίες για να δουν πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι κανόνες θέλουμε υποβολή αναφορών, χρειαζόμαστε τις πληροφορίες, καλύτερη κατανόηση της αγοράς. Δεν θέλουμε να έχουμε δεύτερη οδηγία για διαθωτικά μέτρα. Θέλουμε να δούμε ε, ποιες διαδικασίες είναι για όλους. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη-μέλη και Κοινοβούλιο. Αυτό θέλουμε. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα που θέλω να θίξω. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια από τις συζητήσεις. Μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία μέχρι το, το τέλος του έτους και όπου μπορούμε να σας βοηθήσουμε, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ γιατί δώσατε απάντηση σε κάποια κρίσιμα θέματα. Πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ εκ νέου τον κύριο Ταραμπέλα για το έγγραφο εργασίας έχει αξία όσον αφορά τη διοργάνωση της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που καταβάλατε. Θέλετε να αναφερθούμε στο χρονοδιάγραμμα ή να το αναφέρω εγώ. Πάρτε λοιπόν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, ξέροντας ότι ο Φιλίπ Ζουβέν θα πρέπει να μιλήσει, πρέπει όμως να μιλήσω γιατί μετέθησαν ε, ερωτήσεις και θέλω να απαντήσω επιγραμματικά. Καταρχάς, για τους σκιώδεις ηγητές, και ο κύριο Έγγελ και ο κύριο Χατζημαρκάκη και εσεί και η κυρία Ρούλα αναφέρθηκαν σε ένα θέμα τη υπεργολαβία. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τι διαδικασίε, και αυτό που είπε και η Γκέφχαρτ θέλουμε οι κανόνε που ισχύουν για τον πρώτο ανάδοχο να ισχύει και για του οποίου ανατίθεται η υπεργολαβία. Και όταν υπάρχει εδοχική υπεργολαβία, είναι αναπόφευκτο να βλέπουμε παρεκκλήσει που πολύ συχνά είναι κακές όσον αφορά εκείνους που εργάζονται και το έργο. Οι δημόσιες προμήθειες δεν θα πρέπει να μην ελέγχονται από τις δημόσιες Μέσω της νέας οδηγίας μπορούμε να οδηγούμε σε σεβασμό των συνθήκων εργασίας. Και η διαδοχική υπεργολαβία πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πάντα υπονομεύει τις κοινωνικές συνθήκες εργασίας. Η κυρία Μπίλτα έθεσε ένα ερώτημα. Ευάλωτες ομάδες. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω ένα σημείο που διαφωνώ. Τα κοινωνικά κριτήρια λέτε ότι τα συμπεριλαμβάνετε στο μέγιστο βαθμό. Όχι, στο ελάχιστο τα συμπεριλάβατε τα περιβαλλοντικά κριτήρια, συμφωνώ, είναι πιο εύκολο να το κάνετε. Βασίζεστε στην ετικετοθεσία κλπ. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, μιλάτε για του ανθρώπου με αναπηρία. Εντάξει, αυτό το ενθαρρύνω και το δέχομαι. Πρέπει να προχωρήσουμε ίσω παραπέρα και τα ευάλωτα άτομα. που είναι μακριά από τον τόπο εργασία ε, που δεν έχουν πάρα πολλά προσόντα και αυτά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Ο κύριος διαδικασία που είναι η πιο οικονομικά θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στην τιμή. Μετά από συζητήσεις με τους συναδέλφους νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ικανοποιητική λύση. Κύριε Σβάμπ, δεν ήθελα να υπονομήσω εσωτερική αγορά μέσω των κοινωνικών συνθήκων και της ταυτοποίησης. 19% του ΑΕΠ είναι οι δημόσιες προμήθειες. δεν καλύπτει το πεδίο εφαρμογή όμω το 19%, 4%. Αν αυξήσουμε το κατόφλιο, είπατε θα είναι ακόμα χαμηλότερη κάλυψη. Δεν θα επισέδω σε λεπτομέρειε. Θα ξανακουβεντιάσουμε. Ετέσαι και άλλε ερωτήσει, χρονοδιάγραμμα. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Έγινε. Δεύτερη, στι 19 Μαρτίου, από ό,τι θυμάμαι, ανταλλαγή απόψεων. Ακρόαση στην Επιτροπή αυτή. 20 Μαρτίου. Νομίζω 20 Μαρτίου το απόγευμα αντί 21 όπω προβλεπόταν αρχικά. Το σχέδιο εκθέσεω ότι διαβιβάσω προς μετάφραση 18 Απριλίου, το αργότερο, άντε και 17 μπορεί. Συζήτηση το σχέδιο εκθέσεως θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες φαντάζομαι για να έτοιμο της 8 Μαΐου. Αυτή είναι η αρχή περίοδου υποβολής τροπολογιών και αυτό είναι ασυνήθιστο. Από 8 Μαΐου μέχρι 8 Ιουνίου στις 12 έχετε χρόνο να υποβάλλετε τροπολογίες ένα μήνα. 11-12 Ιουλίου και 6 Σεπτεμβρίου, διότι έχουμε θερινές διακοπές που παρεμβάλλονται, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες σε δύο φάσεις. Για τις συμβαστικές τροπολογίες 17-18 Σεπτεμβρίου 2012, άρα μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο εκθέσεως στην ΙΜΚΟ στην Επιτροπή μας 10 Οκτωβρίου και λογικός, αν όλα πάνε καλά, θα δούμε τι θα κάνει και το Συμβούλιο, θα γίνει τι διαπραγματεύσει. Αλλά με τι συστάδε, με τι ομάδε προτάσεων κλπ. μπορούμε να προχωρήσουμε καλά και να κάνουμε σωστή ανταλλαγή απόψε με το Συμβούλιο και έτσι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο από 10 μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν έχω να πω κύριε Πρόεδρε. Right. Well, thank you very much indeed. Uh, just to confirm from our side, um... Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε συμφωνήσει ότι στις 20 του μηνός θα γίνει η ακρόαση ε, και για τις δημόσιες συμβάσεις 31 το πρωί, από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε δώσει και στο χρονοδιάγραμμά μας πάρα πολλές ευκαιρίες για τροπολογίες, για συμβιβαστικές τροπολογίες, οπότε ελπίζω όλοι να νιώθετε ότι είναι μια πάρα πολύ πλήρης και διεξοδική εξέταση του θέματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλος ιδιαίτερο τον εισηγητή. Τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη εξίσου σημαντική πρόταση που έχει σχέση με αυτό που συζητούμε για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης. Ο Φιλίπ Ζουβά είναι ο εισηγητή μας. Τόση ώρα μας παρακολουθεί προσεκτικά. Βλέπω ότι έρχεται και ο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Οπότε θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Είναι εδώ η σκιώδης εισηγητή, Μπουζόη, Πενσέρι, Ρούλε, Νίκ. και εγώ βεβαίως, ο κύριος Ντεγιόγκ, δεν ξέρω αν ο κύριος Αλβίν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει θα ακούσουμε μια σειρά παρεμβάσεων από τους σκιώδεις εισηγητές και μετά θα δούμε πόσο χρόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε στους ομιλητές μας. Και βέβαια θα δώσω, και το ρόλο στην θα δώσω το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον κύριο Ζουβέν για να συνοψίσει. Κύριε Ζουβέν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγγραφο εργασίας, που είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης και σας δίνω το λόγο να μας το παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με έναν έκδοτο. Με επισκέφθηκε μια επιχείρηση πριν από μερικέ εβδομάδε, πολύ μεγάλη επιχείρηση, γαλλική, που μου που θα μου δώσει τη δυνατότητα να, έτσι, να πω λίγο ε, μερικά πράγματα για εκείνη και θα, μέσω εκείνης θα πω και ορισμένα ε, πολύ κακά πράγματα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σε πολύ λίγη ώρα κατάλαβα ότι όταν μου μιλούσε, μιλούσε για αυτό το θέμα, για το, την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι σύμβαση παραχώρησης και τι δεν είναι. Αυτή είναι η πρώτη προκατακτική μου παρατήρηση. Εγώ αναρωτήθηκα για την καταλληλότητα ενό τέτοιου κειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά την άποψή μου με του ορισμού απάντησα στο ερώτημα αυτό. Μία από τις βασικές δυσκολίες στην παραχώρηση είναι ότι σε κάθε μία από τις παραχωρήσεις ε, λειτουργούμε βάσει του εθνικού μας δικαίου. Μία παραχώρηση ε, στο, στη Γαλλία δεν είναι παραχώρηση στην Ιταλία, στην Πορτογαλία. Δεν μιλάμε τέλος πάντων για το ίδιο πράγμα σε όλες τις χώρες και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να έχουμε έναν κοινό ορισμό επιτέλους, χωρίς αυτό βέβαια να αλλάζει το νομικό καθεστώς ε, του τι είναι παραχώρηση. <clears throat> Τρίτον, ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες καταστάσεις. Υπάρχουν μεμονωμένες καταστάσεις ορισμένων τομέων δραστηριότητας ορισμένων χωρών που τους ανησυχούν ότι βλέπουν την ε, ανάδυση ενός νέου νομικού καθεστώτος. Και θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν τρόποι να εξετάσουμε με αρκετά συνολικό τρόπο το, τα ύδατα, την ενέργεια, τους λιμένες, ε, τις ε, ε υπηρεσίες ε, καθαρι, οδοκαθαρισμού στις διάφορες χώρες. Τέλος πάντων υπάρχουν διάφορα στοιχεία ανάλογα με τις κατηγορίες για τις οποίες μιλάμε και πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Πρώτα όμως ο ορισμός της παραχώρησης, της σύμβασης παραχώρησης. Ε, έχουμε διαφορετική, διαφορετικό ορισμό. 25 αποφάσεις του δικαστηρίου υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφινιστεί αυτό το θέμα. Ε, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι δημόσια σύμβαση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μία σύμβαση παραχώρησης είναι μία σύμβαση με μία δημόσια αρχή που αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ε, ενός έργου, μιας ε, υπηρεσίας σε μία άλλη εταιρεία. Υπάρχει κάποιο λοιπόν που θα αναλάβει τη δραστηριότητα, κάποιο που θα αναλάβει ένα κίνδυνο, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό δεν υπάρχει παραχώρηση και άρα δεν καλύπτεται από την οδηγία. Και σε πολλές από τις δραστηριότητες που φοβούνται ένα τέτοιο είδο κείμενο πρέπει να δοθούν ε, ε, κάποιες γιατί δεν θέλουν να τι αποδεχθούν. Λοιπόν, Πρέπει να είναι πολύ σαφής ο ορισμός, καταρχάς, και κατά δεύτερον, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί και όχι τόσο στα εκτιμώντας, αλλά στο διατακτικό του κειμένου, ενδεχομένως στο πρώτο άρθρο. Να λέμε ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να ε, ε έχουν την ευχέρεια της επιλογής του τρόπου και του μέσου. Για παράδειγμα, τα τελεφερίκ στην Αυστρία, ένα ζήτημα που έχει προκύψει. Βέβαια τα τελεφερίκ αν θέλουν οι δημόσιες αρχές να διατηρήσουν ε, ε, σε εσωτερικό επίπεδο τη μία ή την άλλη δραστηριότητα ε, πρέπει να είναι δυνατόν. Δεν πρέπει οι δημόσιες αρχές να θεωρούν ότι πρέπει να περάσουν σε μία σύμβαση παραχώρησης υποχρεωτικά. Δεν θέλει αυτό να κάνει το κείμενο, επιτύχει το κείμενο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το λέμε στο άρθρο 1 για να κοιμούνται όλοι ήσυχοι. Λοιπόν, σαφή ορισμό, σαφή ορισμή, Το είπα αυτό ήδη. Τι είναι και τι δεν είναι σύμβαση παραχώρηση. Επίση, να πάρουμε το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλό είναι. Αλλά πρέπει να το αλλάξουμε, να το ελαφρύνουμε με μια φιλοσοφία τη διαφάνεια. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ε, ακόμη χώρες ε, ε, στις οποίες περνάνε στο παρασκήνιο τέλο πάντων κάποιες ε, συμβάσεις. Ε, ξέρουμε τι καταχρήσεις μπορεί να υπάρχουν αν δεν υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να έχουμε κανόνες, αλλά απλούς διαφανείς που δεν περιπλέκουν τη ζωή των δημοσίων αρχών. Τι σημαίνει αυτό? Κανόνες που θα επιβεβαιώσουν ότι κριτήρια που θα έχουν ελεύθερα επιλεγή, οικονομικά, ποιότητα, κοινωνικά, ε, τέλος πάντων αυτό που θα επιλέξει κάθε δημόσια αρχή, ελεύθερα αυτά τα κριτήρια γνωστοποιούνται, δημοσιοποιούνται και οι ιδιωτικές αρχές που θέλουν να ε, ανταποκριθούν θα ανταποκριθούν. Πρέπει να είναι πιο ελαφριά η διαδικασία, λιγότερο περίπλοκη και κατά τη γνώμη μου ε, ε, εξακολουθεί να είναι αρκετά περίπλοκη η όλη διαδικασία. Τώρα, Προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις, ε, καλές είναι αυτές προβλέπονται από το κείμενο, ε, να προσθέσουμε κι άλλες προτείνω εγώ. Για παράδειγμα, μία υπηρεσία βλέπει μία τιμολόγηση που δεν μπορεί να την αλλάξει, την ορίζει το κράτος. Τότε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή, όχι. Άρα, πρέπει να προβλέψουμε κάποιες εξαιρέσεις ε, που θα εξακολουθούν να καθησυχάζουν κάποιους ε, που θα ανταποκριθούν ε, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέτοιου είδους συμβάσεις παρά Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε και να δώσουμε την ελευθερία στις δημόσιες αρχές να διαλέξουν τον τρόπο διαχείρισης της όλης διαδικασίας. Και κάτι ακόμη το οποίο αναφέρεται είναι το θέμα της συνεργασίας δημοσίου με δημόσιο τομέα. Το είπα ήδη πολλές φορές, η δημόσια αρχή πρέπει να διατηρεί την ελευθερία να κάνει την επιλογή της, ειδικότερα όταν βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας δημοσίου με δημόσιο. Μετά μπορούμε να μπούμε βέβαια σε λεπτομέρειε που μπορεί να είναι περίπλοκες μερικέ φορέ, γιατί οι δημόσιε αρχέ μπορεί να χρησιμοποιούν νομικέ οδού ε, που επιτρέπουν τη συμμετοχή την ιδιωτική. Εντάξει, αυτό γίνεται. Αν υπάρχει πολλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κάπω μεταμφιεσμένη επασή περιπτώσει η ιδιωτικοποίηση αλλά τότε τι να κάνουμε τότε. Πρέπει να περάσουμε από την σύμβαση παραχώρηση. Αν είναι ελάχιστη η συμμετοχή αυτή τότε νομίζω ότι μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι δεν καλύπτεται από το καθεστώς της παραχώρησης. Θα ήθελα να δώσω χρόνο στη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συζητηθούν τα θέματα αυτά, αλλά θέλω να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Είμαστε κατά του κειμένου γιατί Θέλουμε στην ουσία να συμμετείχουμε καθένα στη γωνίτσα του, να κάνει τα δικά του. Α, ναι, θα σου δώσω εγώ μια σύμβαση, μεταξύ μας, θα τα κανονίσουμε κλπ. Αλλά να το πούμε για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας τότε. Ε, και τότε δεν θα εγκρίνουμε το κείμενο, δεν θα συμφωνήσουμε το κείμενο. Αν όμως φοβόμαστε το, την, το, τη γραφειοκρατία, Εντάξει, αυτό το δέχομαι, πρέπει να πάρουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να το επεξεργαστούμε, να το ελαφρύνουμε, για να είναι χρήσιμο τέλος πάντων. Και πάση περιπτώσει, α μην γελιόμαστε αν υπάρχει κανόνα, ε, ε, ε, πρέπει να ακολουθείτε. Αν θέλουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις ε, ε συμβάσεις, πρέπει να έχουμε κανόνες. η διαφθορά στη χώρα μου ήταν τεράστια μάστιγα. Πριν από χρόνια υπήρχε ε, μια τεράστια υπόθεση που αφορούσε δημόσιες συμβάσεις ε, για, σε διάφορες πόλεις, μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Υπήρχαν τότε κάποιοι κανόνες που εισήχθησαν, έξυπνοι κανόνες, ε, διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια, αλλά άφηναν τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να πούν σε διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση η οποία ουσιαστικά δεν ε, έθετε να αμφιβόλω κανένα απολύτως δικαίωμα από κανέναν. Τι να σας πω, ε, δεν συμφωνώ βέβαια με το να μην προχωρήσει το κείμενο αυτό, γιατί τότε θα παραμείνουμε στη ζούγκλα που είμαστε σήμερα και καμιά φορά, ξέρετε, στη ζούγκλα μπορεί να δούμε και κανένα λιοντάρι και να μην μας αρέσει. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να αποσαφηνίσουμε το τι θα πει σύμβαση παραχώρηση καταρχά. Και αυτό νομίζω ότι ήδη θα καθησυχάσει πάρα πολύ κόσμο και θα διασκεδάσει πάρα πολλέ από τι ανησυχίε που υπάρχουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για η σαφή εξήγηση. Πολύ καλά τονίσατε τα βασικά προσυζήτηση σημεία. Να δούμε τι έχουν να πούνε σκιώδει. Ο κ. Παντζέρη και ο κ. Μπουζόη μετά. Ο κ. Παντζέρη πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ενθαρρύνω εγώ τον κύριο Ιουβέν διότι ε, διερωτή κατά πόσο έπρεπε να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό διερωτώμενα αν έπρεπε να ρυθμίσουμε το θέμα της ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρηση. Είναι καλό το έγγραφο, καλύπτει θέματα που αναφέρθηκαν σε διάφορες ε, συναντήσεις που διεξήχθησαν και αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Η προστιθέμενη αξία της προτάσεω είναι ποιου κανόνες αναφέρει που χρειαζόμαστε, τα βασικά προβλήματα, την προβληματική και τα συμπεράσματα για τη ρύθμιση των προβλημάτων. Επανειλημμένα αναφέρθηκε ότι υποστηρίζουμε την νομοθετική επιλογή που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει σκοπό όχι τόσο να προωθήσει τις συμβάσεις παραχώρησης αλλά να θέσει σαφές νομικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των συμβάσεων. Εξού και η ανάγκη και η σκοπιμότητα νέας νομοθετικής παρέμβασης διαχωριστής από τις δημόσιες συμβάσεις ε, που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συμβάσεων παραχώρησης. Μετά, συμφωνούμε ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ορισμός ε, σαφής των συμβάσεων παραχώρησης που να μην αντιγράφουν ακριβώς την οδηγία για τις δημοσιοπρομήθειες οι κανόνες υπάρχουν έννοιε ιδιαίτερε που αφορούν τι συμφωνίε παραχώρηση αξίες και όχι τιμή αναδιαπραγμάτευση. Απαιτεί κάποιο βαθμό ευελιξία αυτό. Πιστεύω ότι πέρα από τα κριτήρια που επιβάλλονται από την οδηγία θα πρέπει να προβούμε σε απλουστεύσεις των κανόνων που ρυθμίζουν επαρκώς το θέμα της διαφάνειας, της μη διάκρισης να μην υπονομεύεται όμως η δυνατότητα δημόσιες αρχές να διαπραγματευτούν με κάποια αυτονομία και διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη συμβάση παραχώρηση. Μετά, όσον αφορά τι βασικές προβληματικές αναφέρονται σε μία στο έγγραφο προσυζήτηση που καλύπτουν τις περισσότερες ανησυχίες που αναφέρθηκαν στι διάφορες και συναντήσεις. Πιστεύω ότι η προσέγγιση που παρουσίασε ο εισηγήτης είναι επικοδομητική. Χρειάζεται να αναγνωριστεί η εξουσία αυτοδιοργάνωση των δημοσίων αρχών, να αποκλειστούν τα in-house από το πεδίο εφαρμογή και θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα κριτήρια για την παραχώρηση υπηρεσιών. Το θέμα των επιδόσεων, performance, παραμένουν κάποιες διευκρινήσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή πρέπει να καθοριστεί επακριβώς. Να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες των κοινωνικών υπηρεσιών. Άρα θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία η παραγραφός 10. Ε, μετά, ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη κοινωνικές πτυχές. Πρέπει να αλλάξει το κείμενο για να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα εργασίας και να εξασφαλίζονται ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Η αρχή της ότιμης αντιμετώπισης στον τόπο εργασίας είναι θεμελιώδου σημασίας και η οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων, το δικαίωμα εργασία και προστασία του χώρου εκείνου να, είναι, ε, να υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας στον τόπο εργασίας. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ευθύνης του αναδόχου όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, κοινωνικής προστασίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων, υγείας, ασφαλείας στον τόπο εργασίας και άλλες δύο πτυχές. Πρέπει να αποφύγουμε οι διαδικασίες που επιβάλλονται να αυξάνουν τη γραφειοκρατία και το κόστος, αδικαιολογήτως. Μπορούν οι αρχές να μπορούν να εξαιρέσουν κάποιους ψηφίους, αν έχουν καταδικαστεί για μια συμμετοχή σε, οργα... σε εγκληματική οργάνωση, έχουν διαπράξει απάτη κλπ κάποια τα ε, να μην σέβονται κοινωνικούς κανόνες, πληρωμές κλπ. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών διασυνοριακό αφορμώντας τις διάφορες παρατυπίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό ενός υποψηφίου. Αυτά τα αιτήματα και σκέψεις εκφράζουμε στον συγητή για να λάβει υπόψη. Τον ενθαρρύνουμε όμως την προσέγγιση του. Πρέπει να προωθηθεί η πρόταση. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο όσον αφορά ε, σύμβαση σε αυτές ε, παραχωρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μπουσόη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, περιεκτικότατη δουλειά του και το έγγραφο εργασία του. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εργάστηκε. Νομίζω ότι θέτει τα σωστά ζητήματα και επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ καλή βάση για τη συζήτησή μας τους ερχόμενους μήνες. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι κάθε άλλο παρατέλειο είναι το κείμενο. Πρέπει να το βελτιώσουμε συζητώντας ε, λεπτομερώς την ουσία τους και όχι μόνο να κάνουμε μια λογική συζήτηση κατά πόσο θέλουμε μια ξεχωριστή συζήτηση ε, για τις ε, συμβάσεις παραχώρησης. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αιτιολόγηση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης για τα έργα, αλλά όχι για τις υπηρεσίες, ειδικό όταν ε, ε, έχει υπάρξει διαφορετική ερμηνεία των ορισμών με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις στο δικαστήριο. Η αποσαφήνιση της, ε, του όρου της σύμβασης παραχώρησης είναι πάρα πολύ σημαντική για να, προ, να επιτρέπει το κείμενο ε, ασφάλεια δικαίου για τις ε, δημόσιες αρχές αλλά και για τις εταιρείες. Είναι σημαντικό αυτό για να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης όπως επίσης και μεταξύ των συμβάσεων για έργα ή για υπηρεσίες. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, τις συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Ε, με απασχολούν κάποια ποσοστά που αναφέρθηκαν, για παράδειγμα το 90% των δραστηριοτήτων ε, που το νομικό πρόσωπο ε, πρέπει να υλοποιήσει στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύμβασης δεν έχω καταλάβει πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε αυτό το, τον αριθμό πρέπει να συμφωνήσω με όσους επέκριναν ε, την αξιολόγηση αντικτύπου, αν κάτι τέτοιο έλεγε η αξιολόγηση αντικτύπου και όσον αφορά ε, την ε, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, καταλαβαίνω αυτά που λέει ο εισηγητής και είμαι έτοιμος να συζητήσω επ' αυτού. Δεν πιστεύω ότι, ότι, ότι η ιδιωτική συμμετοχή πρέπει να καθορίσει τα πράγματα γιατί μπορεί να είναι ε, η, μειοψηφία. Ε, νομίζω ότι η επιλογή πρέπει να επαφίεται στην, ε, στο νομικό ε, πρόσωπο. Νομίζω ότι σε σχέση με τις συνδεδεμένες ή μη συνδεδεμένες ε, επιχειρήσεις, ε, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι επίσης ε, τα κριτήρια του έργου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, δεν πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, γιατί δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και με τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, τώρα, το να μην σχετίζεται με το, με το θέμα, με, την, με το αντικείμενο του έργου, δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Για, νομίζω όμως ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Και για να, το, να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι έχουμε κάποια εμπειρία σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις που τις συζητήσαμε και είναι, είναι χρήσιμο να τη λάβουμε υπόψη παρά το γεγονός ότι η δημόσια σύμβαση είναι κάτι διαφορετικό από τη σύμβαση παραχώρησης. Μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας στο παρελθόν με τις δημόσιες συμβάσεις και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ε, σε σχέση με τις συμβάσεις παραχώρησης και το σχεδιασμό ενός συνόλου κανόνων που θα είναι εποφελές και επικερδές και για τις εταιρείες αλλά και για τις δημόσιες αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θέλω να το μετατρέψω σε ιδεολογική συζήτηση, ούτε εγώ θέλω κάτι τέτοιο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εισηγητής στην αρχή ότι χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό διότι η παραχώρηση, λέξη παραχώρηση σημαίνει διαφορετικά πράγματα στις διάφορες χώρες. Όπως είπατε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ορισμός που δεν επηρεάζει α, τις νομικές διευθυντές στα κράτη-μέλη ούτε δημιουργεί νέο γραφειοκρατικό άκθος. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες ε, παραχωρήσεις όπως στον τομέα των υπηρεσιών ε, που διαφέρουν από τις άλλες παραχωρήσεις, κυρίως όταν μιλάμε για κοινοφελείς ε, υπηρεσίες κοινού οικονομικού συμφέροντος. Μιλάμε για μεταφορά καθηκόντων που είναι κυβερνητικά καθήκοντα σε άλλο φορέα, σε άλλο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ διαφορετική ρύθμιση διαφορετικοί κανόνες από αυτούς που υπάρχουν για την αγορά προϊόντων ή αγαθών ε, που χρειάζεται διαφορετική δομή, πολύ διαφορετική. Γι' αυτό λυπούμε διότι η μελέτη αντιχτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρειάζεται νέα μελέτη ε, αντιχτύπου γιατί χρειαζόμαστε ε, συζήτηση για το ποιοι κανόνες θα ήταν χρήσιμοι στον τομέα, ποιοι είναι οι κανόνες θα ήταν χρήσιμοι. Όχι να πάρουμε διατάξεις από άλλο τομέα για να εφαρμόσουμε σε αυτό το περιπλοκότατο τομέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν βρείτε λύση καλά και άγια, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι κανόνες θέλουμε. Χρειάζεται να βρεθεί ένα σαφής ορισμός του τομέα και τι θα κάνουμε με τις κοινοφελείς οικονομικές υπηρεσίες. Παράδειγμα, νερό. Αν αναθέσεις την ευθύνη για, τη, για τα υγρά απόβλητα, για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων την αναθέσεις κάπου, ε, βάζεις πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους άλλου άλλου είδους προσέγγιση σε αυτό το τομέα πρέπει να ακολουθηθεί από ότι για κάτι πιο εμπορικό. Το άρθρο 11 είναι περίπλοκο και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη νομική ανασφάλεια από ό,τι αναφερεθεί το άρθρο. Δεν είμαι υπεραφερές σε αυτού. Όσον αφορά τη σύμπραξη δημοσίου-δημοσίου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά πόσο αυτός ο τομέας θα πρέπει να ανοίξει και για τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει γνωμοδοτήσει από αυτού, έχει πάρει απόφαση και γενικά δεν θα πρέπει να αυξάνουμε τη νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τις συμπράξεις αυτές. Ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτει η οδηγία. Όταν μιλάμε για υπηρεσίες, μιλάμε για ένα τεράστιο τομέα. Πρέπει να καθορίσουμε ποιες υπηρεσίες στην Ευρώπη μπορούν να καλύπτονται από κάποια ρύθμιση και ποιες θα πρέπει να μείνουν εκτός. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι εάν αποφασίσουμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους ρύθμιση όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει για τις καθολικές δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινοφελείς υπηρεσίες και δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Um, ε, από κοινού σκιώδη εισηγητή, θα ήθελα και εγώ να πω ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων. Να πω όμως και μερικά ακόμα. Το κριτήριο ανάθεση, ειδικότερα στη σύμβαση παραχώρηση, θα είναι πολύ πιο δύσκολα και περίπλοκα λόγω τη φύση τη πρόταση. Νομίζω όμω ότι πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Για μένα αυτό ε, είναι μεγάλη σημασία. Όσον αφορά τώρα τα πιο μακροχρόνια συμβόλαια, Δύο πράγματα. Πρώτον, πιστεύω ότι η επίδοση, οι ε, ε, των υπηρεσιών είναι ένα απόλυτο κριτήριο Δηλαδή, οποιοδήποτε αναθέτει κάτι τέτοιο θα ήθελε να συμπεριλαμβάνεται στην σύμβαση. Ε, υπάρχουν λοιπόν βασικές, βασικά κριτήρια επίδοσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει επίσης να δούμε και τι μοντέλο εσόδων έχει προβλεφθεί στη σύμβαση. Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση της ε, σύμβασης, μπορεί να υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις των κριτηρίων, ειδικότερα σε περίπτωση μη ικανοποιητική απόδοσης εξωτερικών παραγόντων, όπως ο κόστος, το κόστος ενέργειας, ε, ε, τέλος πάντων κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που πρέπει να τους διαχειριστούμε. Τώρα το ευρύτερο ζήτημα είναι η ειδική φύση οι ευρύτερες διατάξεις ε, της ε, συνθήκης ε, αλλά και οι διατάξεις της οδηγίας των δημοσίων συμβάσεων κατά πόσο μπορούν από διαδικαστικής απόψεως και από άλλης απόψεως βέβαια να εφαρμοστούν και νομίζω ότι ο κύριος Ζιβέν δίκιο έχει όταν λέει για τα προβλήματα των ορισμών Στη δική μου τη χώρα οι συμβάσεις παραχώρησης ε, την κάνουν διαχείρισης ε, ε, από την ίδια αρχή που διαχειρίζεται και τις δημόσιες συμβάσεις και μέχρι τώρα λειτουργεί εύρυθμα αυτό το σύστημα. Είναι όμω μια εντελώ διαφορετική διαδικασία τώρα και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πρόταση, την οποία την έχουμε και πρέπει να την ε, μεταχειριστούμε με επικοδομητικό τρόπο. Αλλά φαίνεται να υπάρχουν πολλές ε, αβεβαιότητες, πολλή αβεβαιότητα γύρω από αυτή την πρόταση σε σχέση με τις προηγούμενες. Κύριε Ντεγιόν, κύριε στο τελευταίο ε, σκιώδη συζητή και μετά έχω έξι ομιλητέ. Ακόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να είμαι σύντομος. Είχα επαφές με ενώσεις ε, επιχειρηματιών ε, από ολόκληρη τη χώρα μου, την Ολλανδία. Μου είπαν την άποψή τους για αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης. και δεν θα ήθελαν νομοθεσία επ' αυτού του θέματος. Εγώ διαβάζω το έγγραφο εργασίας και για μένα σταματάει στο πρώτο σημείο. Εκεί τελειώνουν όλα κατά τη γνώμη μου. Κανόνες, ε, δημόσιες αρχές, ε, μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Κύριε Ζουβέν, εγώ έχω πάρα πολύ απογοητευτεί. Στη συνεδρίασή μας σε Στρασβούργο μας είπε ότι θα είχε μια πολύ καλή νομική ανάλυση από την ομολογία του δικαστηρίου βλέπω ότι έχετε πάρα, πολλά, πάρα πολλές αφάσεις του δικαστηρίου που αναφέρετε και να σας πω την αλήθεια, το επιχείρημά σας νομίζω ότι μόνο σας το πνίγεται σε ένα σημείο της έκθεσης, του εγγράφου, συγγνώμη. Μας λέτε ότι υπάρχει η επιθυμία της νομοθεσίας αυτής, αλλά νομίζω ότι αξιολόγηση αντικτύπου θα έπρεπε να γίνει. Θα ήθελα να μας πείτε πληροφορίες, βέβαιες πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ομολογία. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι θα φάμε λίγο από το χρόνο του κυρίου Έγγελ, γιατί έξι ομιλητές έχω ακόμη. Πάλι δύο λεπτά ο καθένας. Ε, και θέλω και στην κυρία Σικόφσκα να δώσω το λόγο. Mrs. Mrs. Uh, Δύο λεπτά έκαστος. Κύριε πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα τον εισηγητή μας για το πολύ ανοιχτό πνεύμα αυτής της πρότασης σε όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα δύσκολα σημεία να τα φωτίσει, να τον ευχαριστήσω. Βρίσκω ότι σε πάρα πολλά πράγματα έχει σωστές παρατηρήσεις και προτάσεις και σωστά πράγματα προτείνει. Θα ήθελα ρητά να αναφέρω ότι εμείς φυσικά, συνάδελφε Ντεγιόν, θα προτιμούσαμε όχι από τους εργοδότες των διαφορετικών κρατών αλλά και από τους εργαζόμενους ε, να πούμε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε περισσότερο να βλάψει από ότι να ωφελήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι δεν θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια στην εσωτερική αγορά για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και η ε, πρόταση βασίζεται σε άρθρο της συνθήκης και γι' αυτό πρέπει να απλουστεύει την ενιαία εσωτερική αγορά. Αν αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε ή έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις πρέπει να διαρωτηθούμε αν προσφέρει κάποιες δυνατότητες θετικές η πρόταση. Σε αυτό το σημείο, Πρόεδρε, μια και εμείς είμαστε νομοθέτες και αν όταν υποβάλλει την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σκεφτούμε αν την επιθυμούμε εμεί αυτή την πρόταση και συμφωνούμε. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν επιφυλάξει και εδώ αυτέ θέλω να τι εξετάσουμε. Δεν είμαστε κατά περισσότερη εσωτερική αγορά και κανόνων και κανονισμών, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε τι προσφέρουν αυτοί οι νέοι κανόνε και κανονισμοί. Δεν είναι αθέμητο το ερώτημα και η μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώ, και το λέω ξεκάθαρα, δεν δίνει απαντήσει για όλα αυτά. Και γι' αυτό τον λόγο και θα συνεχίσω την παρέμβασή μου για να μπορέσουν αυτά να, να συνάδουν αυτά που προσφέρει ως σαφείς στόχους διαφάνεια, καταπολέμηση διαφθορά στην εσωτερική αγορά ο κύριος Ζουβά και από την άλλη πλευρά αυτά που απουσιάζουν ως στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων με καλύτερο τρόπο να γνωρίζουμε, με πιο αξιόπιστο τρόπο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Μόνο τότε μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα. Το να πούμε «Α, κάποια προβληματάκια υπάρχουν να κάνουμε μια οδηγία» δεν είναι θεμητό και δεν είναι κάτι σωστό για μα αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι φόβοι που συνδέονται με τις παραχωρήσεις. Θα υπάρχουν περισσότερες ρυθμίσεις, λιγότερη ευελιξία, ιδιαιτερότητα της εσωτερικής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη και το καθεξής. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το κείμενο θα δημιουργεί περισσότερο διοικητικό άκτο ή αν θα ενισχύει την εσωτερική αγορά. Διαβάζοντα την πρόταση βλέπει κανείς ότι οι περισσότερες ε, ανησυχίες καθησυχάζονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ασφαλείας δικαίου. Και αν δείτε τι ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δείτε και τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πάνε σε αντίθετη κατεύθυνση, πραγματικά μπερδεύεται κανεί. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που απαντούν στο ερώτημα του κεντογιών και τη συνολική διάσταση και του διάφορου κινδύνους. Ε, πράγματι δημιουργείται σύγχυση και το μεγαλύτερο πρόβλημα η εσωτερική αγορά είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και η σύγχυση που απορρέει από αυτό. Και αν μιλήσετε με τους διάφορους οικονομικούς ε, ενδιαφερομένους θα το δείτε αυτό. Είμαστε σε μια διεθνή διάσκεψη που αφορά τις ε, παραχωρήσεις αυτές και βρήκα αντίλογο σε κάθε πρόταση που εξέφραζα και φαινόταν ότι καθένα χρησιμοποιούσε τη δική του γλώσσα, τη χώρα του και τους δικούς του ορισμού. Το συμπέρασμα που συνήγαγα ποιο ήταν, ότι η αγορά για τις παραχωρήσεις είναι εντελώ κλειστή ακόμα και σε εσωτερικό μιας χώρας και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και αν διαβάσετε τις προτάσεις, οι περισσότεροι φόβοι καθησυχάζονται από το έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, το πεδίο εφαρμογή κλπ. Αν διαβάσετε την, το θέμα της συνεργασίας, εμείς πρέπει να διευκρινίσουμε το θέμα. Δεν θα έχουμε καλύτερη αξιολόγηση επιπτώσεων. Θέλω μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη σαφήνεια, ε, πιο εύκαμπτη προσέγγιση. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο. Δεν πρέπει να κολλήσουμε στου φόβου μα στην αρχή. Αυτή είναι η δουλειά μα, να κάνουμε τη δουλειά μα. Γιατί αν δεν είμαστε ακριβεί και αν επικρατήσει μεγαλύτερη σύγχυση από ό,τι τώρα, δεν θα έχουμε πραγματική εσωτερική αγορά στον τομέα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά το τελεφερίκ όταν κάποιος αναφέρθηκε στην περιορισμένη συνολική διάσταση. Μιλάμε για τον αριθμό των τουριστών που πηγαίνει σε έναν τόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε όσον αφορά τη νομική αβεβαιότητα και νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Thank you. Uh, next, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Γκέπχαρτ. Yeah, Η κυρία Γκέπχαρτ, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εμείς πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουμε και τα αποτελέσματά του σίγουρα είναι θετικά υπό το πρίσμα των σοσιαλδημοκρατών θεωρούμε σωστά αυτά στις πτυχές τους και θέμητα και πολλοί λένε ε, δεν χρειαζόταν να γίνει τίποτα άλλο όμως μια και έχουμε μεγάλο αριθμό αποφάσεων που προέρχονται από το δέκτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που θα συνεχίσουν να έχουμε, θα συνεχίσουν αυτές οι αποφάσεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη εδώ να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα ως Ευρωβουλή και να μην τα αφήνουμε αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίζει τι θα γίνεται στο πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό η δική μου ομάδα δεν είχε ποτέ αμφιβολίες, δεν άφησε ποτέ αμφιβολίες στο να λέμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια οδηγία, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σαφήνειας και διαφάνειας. Η ομάδα μας όμως ποτέ δεν είπε ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνεί. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος και πολύ προσεκτικά όσον αφορά την ουσία της πρότασης. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Ζουβέν για την προσέγγιση του και τον ευχαριστώ πολύ, διότι ακριβώς αυτά τα προβλήματα κατέδειξε που αφορούν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακριβώς όπως και ο σκιώδης εισηγητής κύριος Παντσέρη το έκανε και υπέβαλε προτάσεις. Το ένα θέμα λοιπόν είναι πράγματι το θέμα των ορισμών και όρων. Και θα έλεγα η πρόταση που υποβάλλεται κύριε Ζούβα στο άρθρο 1 να υπάρξει αυτή η αποσαφήνιση, η διευκρίνηση <clears throat> ότι σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και των ρυθμίσεων των αδειών αυτών αλλά για διαφάνεια να μεριμνήσουμε να υπάρξει διαφάνεια είναι μια πολύ καλή πρόταση αυτή θα έλεγα επίσης ότι και κάποια άλλα θέματα διατυπώνεται που είναι πολύ σημαντικά και αυτά η ομάδα μου πάντα επανειλημμένα έλεγε ότι είναι σωστό και σημαντικό αυτά που αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για τέτοιου είδους άδειες να λαμβάνονται υπόψη και να ισχύουν πάντα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κριτήρια υποβάλλει και δυσχεραίνεται αυτό το πλαίσιο. Και αυτό είναι θεμητό ερώτημα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα έλεγα όχι. Παραμένουμε στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και διαγράφουμε αυτά τα πρόσθετα κριτήρια. Για το επιπλέον ερώτημα που πρέπει να διατυπώσουμε είναι ποιοι τομείς καλύπτονται σε σχέση με αυτές τις ε, εγκρίσει άδειε και μπορεί η οδηγία έτσι να λειτουργήσει. Βλέπω κάποιες κάποια μηνύματα να συντομεύσω και να ολοκληρώσω και θα υποβάλω μία πρόταση τώρα μόνο γιατί άκουσα πως έχει η συζήτηση και ο κύριος Ζουμέ έθεσε αυτό το ερώτημα στην αρχή της παρεμβασή του θα έπρεπε πρώτα απ' όλα στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να αποσαφηνίσουμε πώς πιστεύει η πλειοψηφία των μελών είναι υπέρ ή κατά μιας πρότασης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρχει σαφής πλειοψηφία για κάτι τέτοιο, πράγμα το οποίο δεν θα ευχόμουν, ε, το ότι δεν χρειαζόμαστε δηλαδή περαιτέρω οδηγία, τότε θα μπορούσαμε να σταματήσουμε το έργο αυτό. Θα ήταν περιττό και θα αναφερόμαστε σε αυτό που είπε ο κύριος Ζουβέν και θα έδινε πίσω, θα επέστρεφε την εντολή του. Αν όμως η πλειοψηφία πει να εργαστούμε επ' αυτού, τότε να συνεργαστούμε επικοδομητικά, να έχουμε ένα καλό κείμενο. Το πρώτο ερώτημα όμως πρώτα πρέπει να αποσαφινιστεί. Ευχαριστώ. Uh, ε, Καλνιέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Φιλίπ Ζουβέ για ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο εργασίας ε, για τις ε, συζητήσεις μας. Ε, συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που βλέπουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπερβολικά περίπλοκη και πιστεύω, πιστεύω ότι μπορούμε να την απλοποιήσουμε, να την καταστήσουμε σαφέστερη και διαφανέστερη. Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου έχουμε επεξεργαστεί η νομοθεσία σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν λειτουργεί κανένα λόγω έλλειψη διαφάνεια ε, και. Ε, ε διακανονισμών που γίνονται μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα εκ των προτέρων. Γι' αυτό είμαι υπέρ ισχυρών και σαφών κανόνων που θα απομακρύνουν τη διαφθορά που υπάρχει σε ε, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις τροπολογίες. Υπάρχει όμως μία ακόμη διάσταση ε, που θα ήθελα να θίξω, την παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2009 έχει περιορίσει την υλοποίηση νέων συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα και δίνει, επιτρέπει μόνο ε, την ε, ύπαρξη συμβάσεων ε, μη ανάληψης κινδύνου από το κράτος και στη χώρα μου αυτό είναι ένα πάρα πολύ περιοριστικό μέτρο γιατί για την κυβέρνηση της Λετωνίας ε, μετά την κρίση είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, διαθέσει ε, κονδύλια για την υλοποίηση των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάη. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ οργανωτικά για την ακρόαση σε κάτι. Είδα το ηλεκτρονικό μήνυμα, Πρόεδρε, ότι η ακρόαση αυτή στις 20 και 21 του μήνα θα διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο στις 21 θα έχουμε τα θέματα υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών και μετά το θέμα των συμβάσεων. Τώρα το είπατε ανάποδα εσείς. Αυτό θα ήταν πρόβλημα για μένα. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση αν γίνεται. Θα ήθελα να σας ξαναρωτήσω, άλλαξε κάτι στον προγραμματισμό και τι είναι αυτό, διότι δεν το προέβλεπα αυτό σε σχέση με την 21η Τρίτου, 21η Μαρτίου και προτάσεις για ε, ομιλητές θα είχαμε. Μια και έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους ε, ε ομιλητές ε, που έχουν προσκληθεί και είχαμε καλή συζήτηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και με τους Δήμους και κοινότητες από τη Γερμανία και θα ήταν καλό να συμμετάσχουν και από πλευρά μα κάποιοι ομιλητέ σε αυτό το σεμινάριο, σε αυτή την ακρόαση. Τώρα για το θέμα τη ουσία. Εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα για μένα. Χρειαζόμαστε ναι ή όχι αυτή την πρόταση. Αναφέρεται χρειάζεται μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και βεβαιότητα, μεγαλύτερο ανταγωνισμό, να είμαστε πιο οικονομικοί στη χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων και πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να επαναλάβω όμω η απόδειξη όλων αυτών με τη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το έγγραφο εργασία, συνάδελφε ε, ε, Ζουβέν που καταβάλλεται προσπάθειες με πολλούς ορισμούς. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα που υπάρχουν και δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί είναι αναγκαία αυτή η οδηγία και τι χρειάζεται από κανόνες και κανονισμούς και πώς θα μπορούσε αυτό το ρυθμιστικό έργο να διαμορφωθεί. Για να δώσω συνέχεια λοιπόν σε αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος Γκέπχαρτ πιο πριν. Θα ήθελα να πω ότι θα επιθυμούσα και την έχουμε τη δυνατότητα αυτή ως κοινοβούλιο και το ανέφερε ο συνάδελφος Σβάμπ αυτό να έχουμε μια impact assessment από πλευρά του Κοινοβουλίου, μελέτη επιπτώσεων, όπου αυτά τα θέματα θα πρέπει να απαντηθούν και να ρυθμιστούν. Διότι πιστεύω πάλι ότι δεν έχουμε επαρκεί απαντήσει. Η impact assessment μπορεί να εξετάσει πού υπάρχει ανάγκη ρύθμισης και κυρίω να δούμε τι προσφέρουν ω αποτέλεσμα χειροπιαστό, ω πρόσθετη αξία αυτέ οι ρυθμίσει. αν προσφέρουν κάτι. Αναφέρθηκε δυσκολία να υπάρχουν ενιαίοι ορισμοί και ορολογία. Είναι δύσκολο για τα κράτη-μέλη και γι' αυτό είναι δύσκολο και οι κανονισμοί δεν έχουμε ένα κενό χώρο εδώ. Υπάρχουν κάποια θέματα που ε, ρυθμίζονται και αφορούν και το θέμα διαφάνειας που θέλουμε να διασφαλίζεται. Τώρα, για εξαιρέσεις και όσον αφορά τις τιμές κατόφλια και για όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν σε σχέση με τις ε, ε, εντολές και τις συμβάσεις. Όλα αυτά θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να τα εκμεταλλευτούμε για να δημιουργήσει σαφήνεια. Ευχαριστώ. Well, Κοιτάξτε, αν θέλετε περισσότερε εργασίε, ε, ο εισηγητή και οι σκιώδε εισηγητέ, ευχαρίστω να το σκεφτούμε. Κυρία Βερνιό, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έγγραφο εργασία. Θα πάω γρήγορα γιατί πιστεύω ότι για το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 25 αποφάσεις του δικαστηρίου. Συμφωνώ με αυτά που είπε και με την άποψη της κυρίας Γκέπχαρτ. Ε, υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ένα κείμενο ε, που να δημιουργεί ασφάλεια ε, δικαίου. Πιστεύω λοιπόν ότι το κείμενο των 83 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στην υπόσχεσή της να μας παράσχει ένα κείμενο που προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Και όπως λέει και το έγγραφο εργασίας, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, γιατί η κατάσταση είναι λίγο αόριστη σε σχέση με τους ορισμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στους ορισμούς αυτούς. Θα ήθελα μόνο δύο προβλήματα να θίξω. Πρώτον, το θέμα της ενέργειας. Καταλαβαίνω τα ερωτήματα σε σχέση με τις ε, εξαιρέσει ε, για την ε, προμήθεια, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα στο άρθρο 8.1 σε σχέση με την διανομή τη ενέργεια γιατί υπάρχει μία ε, γιατί μία σύμβαση που ανα, ε, ανατίθεται σε μία ε, αρχή ε, διαχειριστική δημιουργεί ένα πρόβλημα για, τους, ε, για τις εξαιρέσεις αυτές. Και αυτό με φέρνει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οριζόντια η εγκάρσια, η οποία μου φαίνεται πολύ πιο περιοριστική σε σχέση με αυτή που προβλέπει ο Ευρωπαίος Δικαστής ε, και αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε στην αυτοοργάνωση και την αυθαιρεσία με την οποία βεβαίως δεν συμφωνώ και όπως λέει και το έγγραφο εργασίας και πάλι συμφωνώ, υπερβάλλουν ζήλος από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, εγγυήσει διαδικαστικέ, ε, ε, περίπλοκα πράγματα, χρονοβόρα και νομίζω ότι βασιζόμαστε στο μοντέλο των δημοσίων συμβάσεων και αυτό δεν ταιριάζει με το καθεστώ των παραχωρήσεων. Είμαι ικανοποιημένη αν μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο της ανασφάλειας δικαίου με ένα κείμενο αλλά, ε, όπως είπε και σε πολλές και πολύ δικαιολογημένες παρατηρήσεις του κύριο Ζουβέν, πρέπει να ανακουφίσουμε λίγο το κείμενο, να το αλαφρύνουμε για να υπάρχει ασφάλεια για όλους τους φορείς, γιατί ε, δεν, ε, δεν είναι καθόλου απλό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σικώσια, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά μπορώ να σας δώσω λίγα λεπτά να μας ε, πείτε έτσι μια προκατακτική άποψη. Αλλά ούτω ή άλλω θα έχουμε χρόνο και τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Μας βοηθούν όλα αυτά για να καταλάβουμε καλύτερα το πώ θα μπορούσε να βελτιωθεί το κείμενο. Θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Θα λάβουμε υπόψη τα όσα υπόθηκαν. Να τονίσω κάτι. Πολλοί διερωτήθηκαν περί τίνος πρόκειται. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται οδηγία. Κάτι θεμελιώδες να πω. Αυτή η οδηγία αφορά ε, το δικαίωμα δικαίωμα υποβάλλει κανείς προσφορά. Δεν έχουμε πληροφορίες δυνατότητα ε, παραχώρησης καθόλου. Δεν έχουμε πληροφορίες όσον αφορά τους οικονομικούς ενδιαφερομένους. Δεν πληροφορούνται όλοι ισότιμα στα κάτι μέλη. Δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές όπως μπορούν για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είναι κάτι που το θυμόμαστε. Πραγματικά αυτή η οδηγία αφορά τη διαφάνεια, αφορά την ισότιμη αντιμετώπιση, τη σαφήνεια και τη βεβαιότητα. Ταυτοχρόνως βοηθούμεθα να αντιμετωπίσουμε πολλά αρνητικά φαινόμενα που εξετέθησαν. Αυτό λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα βαθμός της ρύθμισης είναι κάτι θεμητό ο βαθμός ε, της ε, νομοθέτησης δεν πρέπει να ε, υπολογίζεται σε αριθμό σελίδων γιατί ένας κανονισμός μπορεί να έχει τρεις σελίδες. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι ουσιαστική σημασία για ένα θέμα. Μπορεί να υπάρχει πάντως τρόπος, όντως έχετε δίκιο, να ευθυγραμμίσουμε την νομοθεσία και να απλουστεύσουμε το κείμενο. Να σας επιστήσω την προσοχή στους ορισμούς. δεν είναι μόνο ορισμοί στο άρθρο 2, αλλά συνοδεύεται από πολλά εκτιμώντας που ε, αποσαφηνίζουν περισσότερο τι θα πει σύμβαση παραχώρησης και τι δεν είναι σύμβαση παραχώρησης και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ε, πολλά κράτη-μέλη. Σε σχέση τώρα με τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ένα μόνο σημείο, ε, το ίδιο μοντέλο είναι με την αναθεώρηση για αυτό το θέμα είμαστε 100% σίγουροι, το είπε και το δικαστήριο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί, να θεωρηθεί μια σύμβαση παραχώρησης ως αποκλειστικά σύμπραξη δημοσίου τομέα. Ναι, για τα κριτήρια. Όντω υπάρχουν διάφορα κριτήρια, ευρύτερα, πολύ πιο ευέλικτα από, τις, από αυτά των δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά τώρα ειδικού τομεί, νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσω κάτι σε σχέση με το νερό. Ε, νομίζω ότι οι τομείς ε, πρέπει να ειδωθούν από την οπτική γωνία ε, το του τρόπου με τον οποίο ε, γίνεται η διαχείριση του θέματος σε κάθε χώρα μέλος. Για παράδειγμα, αν ένα κράτος έχει 17 τρόπους να διανέμει το νερό, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο της οδηγίας ε, του, όλους αυτούς τους τρόπους. Όσον αφορά τώρα τα κοινοφελείς υπηρεσίες... Σε αυτέ τι υπηρεσίε αναφέρονται πολλέ αποφάσει του δικαστηρίου, γι' αυτό ακριβώ ε, καλύπτονται. Το κατά πόσο η νομολογία είναι σαφή ή όχι, νομίζω ότι έχουν δοθεί απαντήσει. Γιατί δεν είναι σαφή, σαφή τα πράγματα, γιατί είναι αντιφατικές, ε, αντιφατικές και γιατί ε, δεν έχουν όλες ολοκληρωθεί ακόμα. Καλώς, πάρα πολύ σημαντική ενακτήρια συζήτηση. Ο Φιλίπ Ζουβέν πραγματικά είναι πολύ περισμένος χρονικά. Ίσως σύνοψη πολύ σύντομη να αναφέρει ακροάσεις, χρονοδιάγραμμα κλπ. Άντε ένα δίλεπτο το πολύ να σου δώσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε δύο λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Θα προσπαθήσω να ψήσω. Ακούστε, πρώτα απ' όλα. Χρειάζεται αυτό το κείμενο. Ειλικρινά. ολο ο είπατε το είπε. Είτε είπατε ότι ήταν αναγκαίο ή όχι, είπατε ότι δεν συμφωνούμε όσον αφορά τον ορισμό. Ακόμα και γι' αυτό δικαιολογείται ένα κείμενο. Τουλάχιστον έχουμε ένα κοινό ορισμό. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. γνωρίζετε όπω και εγώ, όταν έχω, σα δούνε κάποιοι σα λένε αυτό το κείμενο δεν μα αρέσει γιατί είναι καλύτερα έτσι που έχουν τα πράγματα και αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι επιχείρημα μεγάλη πολιτική ηθική. Υπάρχουν κάποιε συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτό. Τρίτον, πιστεύω ότι το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περιπλοκότατο. Συνεργάστηκα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο καλός. Το επαναλαμβάνω. Αντίθετα με αυτό που είπαν κάποιοι. Χρειάζεται να υπάρχει κοινό ορισμό, ή πρέπει να επικρατεί διαφάνεια, αλλά θα πρέπει να είναι, να είναι απλούστατα τα πράγματα. Δεν είναι το κείμενο που είναι περίπλοκο μόνο, όλο και περισσότερο και στα, στις χώρες μας βλέπουμε και στα κοινοβούλια μας ότι οι νόμοι γίνονται πιο φλίαροι, περίπλοκοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα κείμενο. Αυτό λέω στην κυρία Κέπχαρτ που λέει ότι ουσιαστικά τι λέει, συμφωνούμε είτε όχι με το κείμενο. Σας λέω απλώ ότι Ε, δεν θέλουμε ένα πολύ αποδυναμωμένο. Εσεί προτείνετε ένα κείμενο πολύ απλουστευμένο, επικεντρώνεται επί του ορισμού, του πεδίου εφαρμογή, τα κριτήρια αναφέρει και μια διαδικασία εξαιρετικά ελαφριά. Και μετά το θέμα της ε, ελεύθερης διατησίας ε, για την τοπική αυτοδίκηση λοιπά. Η κυρία Ρούλε είπε κάτι. Είπε, προσέξτε, μην διαταράξετε το νομικό σύστημα των κρατών μελών. Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Διερωτήθηκα, μήπως για να ξεφύγουμε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο όρο από τον όρο παραχώρηση. Να εφεύρουμε νέο νομικό όρο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε σήμερα. Ότω ώστε εκείνοι που κάνουν τι παραχωρήσει στα κράτη-μέλη να κάνουν δικέ παραχωρήσει και εμεί να έχουμε ένα νέο δικό μα νομικό μέσο. Είναι μια λύση νομίζω ότι χρειάζεται θα ετοιμάσουμε ένα κείμενο πάρα πολύ επιχειρησιακό, λειτουργικό, ελαφρύ, εύκαμπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος μιλάει εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Ζουβέν και ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ο κύριος Ζουβέν σωστά σκέφτεται όπως το βλέπω εγώ το πράγμα, αλλά είναι αρκετά ριζοσπαστική προσέγγιση, άρα προφανώς πρέπει να το συζητήσουμε μαζί σας ε, και τους κοιόδης να δούμε αν χρειάζεται μια εξωτερική άποψη να εκφραστεί. Θα υπάρξει 21 Μαρτίου μια ακρόαση η οποία ίσω να διαφωτίσει το θέμα. Θα πρέπει να οργανώσουμε την ακρόαση να το κάνει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που έχει δημοσιευτεί για την ώρα. Η έκθεση θα πάει μετάφραση 25 Απριλίου. Θα συζητηθεί 29-31 Μαΐου, προθεσμία για τις τροπολογίες 21 Ιουνίου και μετά συζήτηση τροπολογιών το Σεπτέμβριο. Προφανώ, αν υπάρξει περιπλοκότερη πρόταση, ίσω χρειαστεί επανεξέταση του χρονοδιαγράμματο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση. Τι κάνουμε με την αξιολόγηση συνεπειών. Αυτή την πρόταση που ακούστηκε. Εάν κάνει αξιολόγηση συνεπιών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό ίσω να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα, ετοιμάσουμε. Αυτή την έκθεση. Αυτό πρέπει να το συζητήσει με όλου μα ο κύριο Ζουβέν και αν προτείνει δραματικά, κάτι που είναι δραματικά διαφορετικό, ίσως αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και να μας δοθούν και κάποιες απέξω συμβουλές. Ίσως θα πρέπει να επιστρέψει συζήτηση στην ομάδα των σκιωδών εισηγητών και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Η παράλληλα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε και την αξιολόγηση των συνεπιών. Η μονάδα η αρμόδια είναι εδώ, την καλωσορίζω. Έχουμε μονάδα αρμόδια για την ε, αξιολόγηση ε, αντιχτύπου και μπορούμε να τις ε, αναθέσουμε να προβληματιστεί επί του θέματος αυτό. Κύριε Πρόεδρε, λέει και ο Ζουβένι, για τη συμπληρωματική αυτή μελέτη αντιχτύπου δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε. Είμαι αρκετά ε, διστακτικός αφορά την ιδέα. Νομίζω ότι είναι ψευτοκαλή ιδέα. Αλλά συμπληρωματική ε, θα, τέτοια έκθεση θα ήταν πολύ καλή. Ξέραμε ακριβώ ποιο είναι το ερώτημα που τίθεται. Αν λέτε ότι χρειάζεται κοινό ορισμό ότι όχι, εγώ έχω απάντηση ξεκίνησα τη συζήτηση που θα κάνουμε με τους σκιώδεις, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως θέλουμε αξιολόγηση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγηση συνεπιών όσον αφορά την πρόταση σε διάφορες περίκοπες. Μπορούμε να το κάνουμε, διότι είναι δική μας η πρόταση και αν είναι πολύ διαφορετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αν η εξολόγηση συνεπειών δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο περίπλοκο τρόπο και στο πετυχαίνεται ένα πλούστερο, έχουμε λόγο να το κάνουμε. Κύριε Έγκελ, ζητούμε συγγνώμη γιατί και εσεί έχετε εργαστεί επί των κρατικών προμηθειών. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση επί τη εκθέσεώ σα τώρα. Θα σα δώσουμε το λόγο για να κάνετε μια παρουσίαση τη πρότασή σα και αν έχουμε ε, χρόνο θα κάνουμε και ένα πρώτο γύρο συζητήσεω των σκιωδών. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσετε την παρουσίαση της εκθέσεώς σας τώρα το πρωί, παρόλο που δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Καλώς. Πρόεδρε, δοθέντω ότι υπό τι πολλέ περιστάσει δεν θα καταλάβαινα και τον εαυτό μου, προτείνω να το κάνω αυτό από τη στιγμή που όλοι θα αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην αίθουσα ή αν θέλουν να φύγουν. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο, θα αφήσουμε όλου του ενθουσιώδει υπέρμαχου ε, για το θέμα αυτό που ενδιαφέρονται να δούμε ε, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε ποιο παρίσταται. Έχουμε το σκιώδη, του σκιώδου. Ο κ. Κρόιτσμαν είναι εδώ, δεν υπάρχουν πράσινοι. Ο κ. Ντε δεν είναι εδώ. Μόνο δύο σκιώδεις έχετε. Η ομάδα μου δεν έχει διορίσει καν σκιώδη η ομάδα μας είσαι είχε κάθε λόγο για να μην έχει σκιώδη ηγετή. So we're not even going to bother. right. Okay, let's go. Um... Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Όσοι διαβάσατε αυτά που έγραψα, θα παρατηρήσατε ότι προσέγγισα κάπως ελεύθερα το θέμα. Κινήθηκα βάσει ανησυχίες πραγματικής για την εσωτερική αγορά μερει για την εσωτερική αγορά. Δεν θα αναφερθώ στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ελλείψεω χρόνου. Θα αναφερθώ στι γενικέ γραμμέ που ακολούθησα. Πέντε σημεία θα αναφέρω. Και θα πω και τι έκανε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Βασικό στοιχείο, κρίσιμο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά πόσο θα ισχύει για όλη την επικράτεια τη Ένωση. Διότι διαφορετικά δεν αφορά την ενιαία αγορά ενδεχομένως δεν αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης και τη αυτή η περίπτωση πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η πρόταση. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι ισχύει είναι ότι ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για νόμο που εφαρμόζεται σε κάποια ζώνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, είναι προφανέστατο ότι μιλάμε για νέο οικονομικό μέσο που θα πρέπει να αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όχι μόνο για να τροφοδοτεί τον προπολογισμό, αλλά και σε περίπτωση κρίσης να παρέχει και άλλους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη εντός της νέας αγοράς. Και αυτό είναι κάτι που προσπάθησα να προτείνω. Δηλαδή, να το εφαρμόσουμε ταχύτερα από αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα δύο χρόνια πριν εφαρμοστεί αυτό, ίσως να μην πετύχει κανέναν από τους σκοπούς που θέλουμε. Τώρα όσον αφορά τα διάφορα ποσά, πρότεινα να τα, να αντιστρέψουμε. Ίσως να φαίνεται παράξενο για κάποιους, αλλά έχει νόημα για μένα, για τον απλούστατο λόγο, για τους συντελεστές αυτούς, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές που είναι χρήσιμες στην αγορά και κάποιες που δεν είναι. Και υπάρχουν κάποιοι τομείς τεχνογνωσίας σε οικονομικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καλύπτονται συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές που θα πρέπει να προστατευτούν ενώ άλλες δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό όλο ο τομέα επενδυτικών ταμείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλού σκοπού για την προώθηση οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και τα συντεξιατικά ταμεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να φορολογούνται λιγότερο από άλλα παράξενα παράγωγα προϊόντα που πιθανότατα θα προσπαθήσουν να διαφύγουν αν επιβληθεί η αδίποτε φορολόγηση σε αυτά αν το κάνουμε αυτό περιθωριακά, λιγότερο περιθωριακά, αυτό δεν επηρεάζει τα πράγματα πραγματικά. Ενώ τα άλλα στοιχεία θα θέλαμε πραγματικά να παραμείνουν εντός της Ένωσης. Τέλος, κάτι για την επιλογή των νομοθετικών μέσων. Ίσως ο στόχος της εναρμόνισης θα εκπληρωθεί καλύτερα μέσω κανονισμού παρά μέσω οδηγίας. Γι' αυτό στο κείμενό μου Λέγω ότι στην αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται θα κάνει του κειμένου να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο μια οδηγία ως έχει θα εξεπλήρωνε το στόχο της εναρμόνισης ή αν θα ήταν λογικότερο να γίνει η επιλογή ενός κανονισμού στο μέλλον. Τώρα, είδα ότι η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα κείμενο το οποίο βεβαίως δεν αναφέρεται σε αυτά τα θέματα, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Η, δημιουργία, η δημιουργικότητά τους είναι χρονικά περιορισμένη. Μονίμως μάλλον περιορισμένη. Όχι μόνο η δημιουργικότητά τους είναι μονίμως περιορισμένη, αλλά και η ετοιμότητά τους να υπερασπιστούν την αρχή της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής σε όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα καταπέσει αν υπάρχουν ε, άκαμπτες αντιρρήσεις ενός ή δύο κρατών. Αλλά καλύτερα από το να Καλύτερα να έχουμε κάτι που ισχύει, να μην έχουμε κάτι να μην έχουμε τίποτα παρά κάτι που ισχύει μόνο στην Ευρωζώνη, που μάλιστα καταστρέφει ότι έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο. Προσπάθησαν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε μέσα που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό διευρύνει το πεδίο και αυτό είναι σωστό και έχει μεγαλύτερο νόημα όσο ευρύτερος ο τομέας γεωγραφικής εφαρμογής του μέτρου ε, τόσο μεγαλύτερο και το νομικό βάρος, η νομική ισχύ που θα έχει το μέτρο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ που δείχνετε το βαθμό φαντασίας ε, ε, που αναμένεται σε αυτή την Επιτροπή έναντι της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Ο κύριος Ντεκάμπος. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε και την καλή διοργάνωση και να τον συγχαρώ για την εφάνταστη δουλειά και τον ευφυή τρόπο. Και έτσι δεν περιοριζόμαστε όσον αφορά τη φαντασία μας θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι συμφωνώ με κάποιες από τι προτάσεις του που είναι καινοτόμε και διαφωνώ με κάποιες άλλες. Αλλά αυτό αποτελεί μέρος της κανονικής καθημερινής ζωής μας ούτως ή άλλως. Πρώτα απ' όλα εξαίρεση όσον αφορά συνταξιοδοτικά ταμεία και τα όργανα συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητα. Αυτό για ε, για ένα τέλος ενός δεκάτου, ένα ποσοστό ενός δεκάτου του ε, συνολικού. Δεν είναι όμως σαφές ε, ποιο είναι το κέρδος ε, που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτή την εξαίρεση. Και με όλες τις εξαιρέσεις δημιουργούνται ευκαιρίες για να γίνουν κόλπα οικονομικά και να υπεκφύγουν κάποιοι. Μία εξαίρεση πρέπει πάντα πολύ προσεκτικά να αναλύεται στις επιπτώσεις. Μόνο τότε αξίζει να δούμε το κόστος αυτής της εξαίρεσης είναι θετικό ή όχι. Και έχουμε μεγάλες αμφιβολίες εδώ σε αυτό το σημείο. Δεύτερο, για την πρόταση του εισηγητή. Η πρόταση αυτή στοχεύει στο να υπάρξει μία αύξηση, στο να εφαρμοστούν όλα αυτά στα παράγωγα και μία αύξηση 0,01. Ξέρω ότι τα παράγωγα έχουν κακή φήμη. Δεν είναι ε, κάτι το οποίο χαιρετίζουν όλοι. Όμως ε, εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μην ρυθμίζονται όλα αυτά αυθαίρετα πρέπει τα παράγωγα να ρυθμίζονται πάντα σύμφωνα με τις προτάσεις και τα συμπεράσματα φυσικά που υποβάλλονται από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και όπως έχει εκφραστεί εκεί. Όμως τα παράγωγα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δεν δικαιολογείται να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά τον, τα τέλη που θα επιβάλλονται και τους φόρους. Ακόμα και το κόστος των συναλλαγών και της ε, ε όλης αυτής ε, θα πρέπει να απλουστεύουν τα πράγματα και να δούμε αν δικαιολογούνται έτσι αυτά τα τέλη. Είμαι πολύ θετικός όσον αφορά την πρόταση του εισηγητή ώστε αυτό να αρχίσει να ισχύει, να ισχύει το 2013. Και είμαι πολύ θετικός επίσης για την υποκατάσταση του οχήματος οδηγίας με ένα κανονισμό που πρέπει να αντικαταστήσει την οδηγία. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή για να κάνουμε εναρμονισμούς με ενιαία τέλη, κοινά τέλη, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την πρόταση, με αυτή την προσέγγιση του κύριου Έγκελ όσον αφορά τροπολογίες από πλευράς του. Και τέλος, για τον ε, προορισμό των εσόδων του taxation, financial taxation. Η πρόταση του εισηγητή είναι να εντάσσονται στον γενικό προπολογισμό τη Ένωση. Εγώ προφανώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτή την προσέγγιση, Όμω μπορεί να υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ δυνατότητε. Και γι' αυτό συμφωνώ περισσότερο με την θέση τη εισηγήτρια τη ΕΚΟΝ, οικονομική Νομισματικής επιτροπή, ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου που θα ισχύει για αυτή την περίοδο. Συμπεραίνω, σε πολλά σημεία συμφωνώ λοιπόν και ειλικρινά πιστεύω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, εφάνταστη δουλειά ο εισηγητής με καινοτόμες προτάσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν όμως άλλες τροποποιήσεις εδώ που αξίζει να δούμε σε βάθος και δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έμαθα εγώ ότι 75% των τελών και φόρων συναλλαγών θα προερχόντουσαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία. Αν δεν συμπράξει, αν δεν συμμετάσχει η Μεγάλη Βρετανία, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο πια να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Κατανοώ ότι ε, αν δεν θέλει τώρα να μην θέλει η Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τις τράπεζες και τις συναλλαγές κάτι τέτοιο, ε, τότε ποιος θα ε, επομιστεί αυτές τις ε, δαπάνες στο τέλος τέλος και πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ο φόρος συναλλαγής θα πληρώνεται από τους πελάτες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τίποτα άλλο και διαφορετικό από ότι ένα φόρο. Ένα φόρο που θα πληρώνει ο πελάτης θέλουμε να καλύψουμε και να ε, επομιστεί το βάρος ε, η ε, ηλεκτρονική συναλλαγή. Όμως εδώ φοβούνται οι Βρετανοί ότι θα πάνε στην Σιγκαπούρη όλη αυτή η δυνατότητα συναλλαγών με αυτόν τον τρόπο. Θα πάνε στη Σιγκαπούρη. Εκείνοι που θέλουμε να πλήξουμε και να επιβαρύνουμε δεν θα επιβαρυνθούν έτσι. Και οι πελάτες θα υπομίζονται το βάρος. Όταν θέλουμε να έχουμε κονδύλια για τη συνταξιοδότηση για τους ανθρώπους που θα βγουν στη σύνταξη θα χάσουμε πολλά κεφάλαια με αυτόν τον τρόπο. Η ιδέα που έχουν οι Γερμανοί φιλελεύθεροι ε, για την επιβολή τελών δεν είναι και τόσο χαζή. Θέλουμε να κάνουμε κάτι και μετά λέγεται εντάξει αυτά που έχουν οι Βρετανοί θα τα εισαγάγουμε στην Ευρώπη, να ισχύουν στην Ευρώπη. Θα υπάρχει level playing field, θα είναι ισοδίκαιο το πλαίσιο δραστηριοποίησης και έτσι θα αναγκαστούν οι τράπεζες να συνεισφέρουν. Ο συνάδελφος Μάντας έχει σημειώσει επίσης να πω ότι να δούμε μήπως θα πρέπει να αναμείνουμε το impact assessment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβιβάζω την πρότασή του μέχρι ότου αποφασίσουμε εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε. Ναι, Αυτά που θέλουμε με άλλα λόγια και ως φιλελεύθεροι θα μπορούσαμε να δεχόμαστε ίσως εκείνοι οι οποίοι προκάλεσαν την κρίση να συνεισφέρουν από πλευρά τους. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί, θα υπάρξει μετεγκατάσταση. Οι πελάτες θα πληρώνουν στο τέλος τέλος τα σπασμένα. Και αυτό θα είναι επιβάρυνση. Διαρωτώ με, για τις λίγες χώρες ε, του ευρώ θα πρέπει αυτά να τα ε, περιορίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι λαϊκίστικο αυτό, ίσως δημοφιλές ή λαϊκίστικο, αλλά αν δεν δίνει τίποτα ως αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν πετυχαίναμε το στόχο θα έλεγαν όλοι εντάξει έχει νόημα, διότι αυτοί θα έπρεπε να πληρώνουν εκείνοι που θα έπρεπε να συνεισφέρουν. Ναι. Και ε, Παρέμβαση χωρί ε, μικρόφωνο. Ναι, το ανέφερα αυτό και προσπαθώ να το εξηγήσω όλο τον καιρό. Όταν 75% των κονδυλίων από το, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εισέρχονται, το οποίο όμω δεν θα συμμετάσχει, δεν έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Σαφέστατα το είπα αυτό προηγούμενα. Ε, να σκεφτούμε λοιπόν απλά και ξεκάθαρα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα το εισαγάγουν αυτό για να υπάρχει ένα level playing field σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία όπω ισχύουν εκεί τα πράγματα. Και αυτή θα ήταν μια συνεισφορά για να υπάρξουν τέτοια κονδύλια. Κατά τα άλλα έχουμε μεγάλε επιφυλάξει. Αν επιτυγχάνεται ο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώ δεν έχουμε χρόνο να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρέπει να κλείσουμε την πρωινή μα συνεδρίαση. Φρανκ Έγκελ, μήπω θέλει να συνοψίσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος πολύ ουσιαστικών ε, σχολείων καταληκτικών. Ε, θα ήθελα να πω στον κύριο Κρόιτσμαντ το ότι μπορούμε μόνο να αξιολογήσουμε ό,τι έχουμε μπροστά μας. Πολύ ε, καλή ιδέα μπορεί να είναι και μια εναλλακτική προσέγγιση, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική προσέγγιση, οπότε πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Εγώ θα περιμένω εναγωνίως ε, τις τροπολογίες και θα ξαναδούμε το όλο θέμα ε, πολύ πιο διεξοδικά. Μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι έχετε χρόνο για υποβολή τροπολογιών. Μπορείτε να απορρίψετε το όλο κείμενο που από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Κρότσμαν θα ήθελε να το κάνει. 20, 20 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και μέχρι τότε θα δούμε και τις εξελίξεις. Νομίζω ότι δεν βλέπω, να, δεν βλέπω να προχωράμε πολύ με αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως ομοφωνία χρειάζονται τα θέματα τα φορολογικά και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει το θέμα ως έχει. Λοιπόν, κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα επανέλθουμε στις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.